έχει συμβάλει πολύ σημαντικά στην ε, προσαρμογή της αγοράς σε δείκτες ενεργειακής αποδοτικότητας. Έχουμε ήδη προϊόντα καλύτερα από την κατηγορία Α και γι' αυτό πρέπει τώρα να επαναταξινομήσουμε και να επαναταξιολογήσουμε την κλάση Α και την προσαρμόσουμε στα νέα δεδομένα. Επίσης πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η ενεργειακή ταυτότητα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ του καταναλωτή και των λιανοπολιτών. Διότι και οι δύο είναι ενδιαφερόμενοι αυτής της μεγάλης αγοράς και είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο ξεκινήματος, ε, μια σημαντική βάση για τα καταστήματα πώλησης, μια βάση καλής επικοινωνίας με τους καταναλωτές. Γι' αυτό πρέπει να είναι το νέο σύστημα κατανοητό και απλό για τους καταναλωτές. Μας ανησυχεί λίγο ε, ο εξή διάλογος που μπορεί να γίνει στο μέλλον μέσα σε ένα κατάστημα αν ακολουθήσουμε την πρόταση της Κομισιόν. Διότι διαφορετικά προϊόντα θα έχουν διαφορετικές ετικέτες. Λέμε, π.χ. ο καταναλωτής μπαίνει στο μαγαζί, θέλω νέο ψυγείο, πλυντήριο και πλυντήριο πιάτων ποιο προϊόν μου συστήνεται για καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Και ο πολιτή λέει, κοιτάξτε σα ενδιαφέρει η ενεργειακή απόδοση, ίσως θα πρέπει να διαλέξετε το α-40 για ψυγείο, τη τάδε μαρκα η α60 για την, ε, ε, της β μάρκας, για, την, ε, για το πλυντήριο ρούχων και α20 για το πλυντήριο πιάτων κατηγορία C ή κατηγορία D για α πλυντήριο πιάτων πάλι από την άλλη μάρκα. Ε, ε, χάος δηλαδή. Γι' αυτό πιστεύουμε, αν ο καταναλωτής μπει σε ένα κατάστημα, είναι σαν να μπαίνει σε ένα λαβύρινθο, ε, στον οποίο θα χαθεί. Αυτό καταλαβαίνετε, μας στεναχωρεί, διότι όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να αυξήσουμε τη ζήτηση των πιο ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων έτσι ώστε και οι κατασκευαστές να έχουν μια σωστή απόδοση των επενδύσεών τους. Πολλές φορές ελέγχθη λοιπόν ότι το α g σύστημα έχει, θα περάσει μια μεταβατική περίοδο που θα είναι δύσκολη να εξήγηθεί στους καταναλωτές. Πρέπει λοιπόν αυτή η μεταβατική περίοδο να, δυστυχώς να είναι συνεχή, διότι συνεχώς ανανεώνονται οι συσκευές και ο καταναλωτή, καταναλωτής συνέχεια αντιμετωπίζει αυτή τη διαφορετική ταξινόμηση από μία μάρκα σε μία άλλη. Διότι ας πούμε η μία μάρκα έχει την παλιά ταξινόμηση ακόμα, η άλλη όμως σε μεταβατική φάση έχει την καινούρια χρειαζόμαστε τώρα πάνω από 7 ε, κλάσεις, ε, ταξινομήσεις κατηγορίες. Από τεχνικής άποψης δεν νομίζω. Εγώ δεν, ε, δεν πιστεύω ότι από τεχνικής άποψης χρειάζεται να προσθέσουμε περισσότερες από 7 κατηγορίες. Διότι αν λάβουμε υπόψη ότι το eco, τα eco-designs, οι προδιαγραφές του eco-design σιγά σιγά η φάση αυτή φθήνει, είναι φθήνουσα ήδη και θα τελειώσει η σημερινή ταξινόμηση B έως G μετά από ένα χρόνο με το α από πάνω νομίζω ότι θα επαρκεί. Πώς μπορούμε να λύσουμε λοιπόν τη μεταβατική περίοδο. Για να δούμε αν θα την καταλάβουν. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε πολλά και να σχολιάσουμε την μελέτη της Κομισιόν γιατί δεν έχουμε δει ακόμα τα συγκεντρωτικά στοιχεία και τα σχόλια. Αλλά από προηγούμενες μελέτες της Κομισιόν βλέπουμε ότι δεν επιβεβαιώνονται τα συμπεράσματα, τα ευρήματα της Κομισιόν. Η Αυστραλία έχει ένα παρόμοιο πρόβλημα. Κάναν μια έρευνα στους καταναλωτές και σμίκριναν την κλίμακά τους και κάναν μία επαναξιολόγηση, επανασχεδιασμό της κλίμακας την οποία την κατάλαβαν οι καταναλωτές και βάσει μιας άλλης μελέτης αν ε, προσθέσετε μία μερομηνία, μία χρονολογία πάνω στην ετικέτα θα το καταλάβουν οι καταναλωτές. Παραδείγματο χάρη μπορείτε να βάλετε την ε, χρονολογία ισχύω τη ενεργειακή ταυτότητα 09 με 011 όπω βλέπετε εδώ οπότε καταλαβαίνουν οι καταναλωτέ ποια κλάση ισχύει για ποια χρονολογία, ποιο χρονικό διάστημα. Η κυρία Ποδηματά επίση ανέφερε τη μελέτη του Σεν Γκάλεν από το α-20% το οποίο επανέρχεται στο α g. Πιστεύω ότι εάν οι καταναλωτές θέλουν να πάρουν καλύτερες συσκευές και σε μεγαλύτερη τιμή και αν κάνουν την, πάρουν την απόφαση βάσου του A ως G και εν συνεχεία αλλάξουν με τη νέα ετικετοποίηση α-20 ή α-60 δεν καταλαβαίνουν ακριβώς ε, ποια συσκευή πρέπει να διαλέξουν εφόσον είναι διατεθειμένη για καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη τιμή. Επανερχόμενοι στην Αυστραλία πρέπει να πω ότι οι καταναλωτές στην Αυστραλία προτίμησαν την, βασικά την ίδια ταξινόμηση με, πιο συμπυκνωμένη, πιο, ε, ε, πιο ουσιαστική δηλαδή και όχι μία επαναξιολόγηση με περισσότερες κατηγορίες, περισσότερες ε, κλάσεις. Όσο περισσότερο αυξάνουμε την ε, ταυτότητα και τις διάφορες κλίμακες, τόσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται καταναλωτής. Ο χρόνος είναι χρήμα και ο καταναλωτής θέλει γρήγορα να καταλαβαίνει τι γίνεται πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε να προχωρήσουμε γρήγορα γιατί έχουμε φτάσει σε ένα διέξοδο, έχουμε κολλήσει. Ε, και στο eco design πρέπει να αναπτύξουμε νέα μέτρα και να προχωρήσουμε. Οπότε εμείς θα θέλαμε να, αποφασίσουν, να αποφασιστεί γρήγορα ε, το νέο σύστημα και δεδομένου ότι οι ταυτότητες από α έως g δείχνουν, δείχνουν ότι αυτές προτιμάει η καταναλωτή σαφέστατα πιστεύουμε ότι μπορούμε να τις ε, ενημερώνουμε τακτικά και να προτιμήσουμε αυτή την κλίμακα. Ιδίω για το α-20 για, για τα ψυγεία που αποφασίστηκε το Μάιο, ε, εάν αυτό αποφασιστεί δεν θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές ε, ταυτότητες για ίδιες συσκευές με ίδιες αποδόσεις στην αγορά την ίδια στιγμή. Να μην υπάρχει δηλαδή αυτή η επικάλυψη στην αγορά των ιδίων μηχανημάτων με διαφορετική σήμανση. Και βρίσκομαι στα αριστερά της κυρία Ποδηματά. Αν θέλετε να απευθύνετε ερωτήσεις σε μένα. θα είμαι ευτυχή να απαντήσω. Ευχαριστώ. Ε, βλέπουμε ότι είναι διαφορετική αξιολόγηση, δεν συμπίπτουν πάντα τα ευρήματα και έχουμε καλέσει και μια ε, τρίτη κυρία, ε, Έρικα Χόπ. Χόπ, πώς σας λένε, δεν ξέρω από το όνομά σας ακριβώς. Έχετε το λόγο. Ε, um, Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Αποδηματά και την Επιτροπή που μας έδωσε την ευκαιρία να σας μιλήσουμε σήμερα εκ μέρους των μη κυβερνικών οργανώσεων για το περιβάλλον. Λέγομαι Έρικα Χόπ και εργάζομαι για το Action Network έχουμε περίπου 3.000 και μη κυβερνητικέ οργανώσει σχετικά με την αλλαγή του κλίματο. Μιλώ και εξ ονόματο του πλέον τη συναδελφάτσα Άμπιχ και Έντερ Τουλού, όπου πιθανώ δεν έχετε συναντήσει. Όπω και άλλοι είπανε, πρέπει να έχουμε κατά νου γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε. Όλοι οι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί στόχοι σχετίζονται με αυτή την ανάγκη χρήση ενέργεια. Έχουμε ε, καινοτομίε, έχουμε πολλέ νέε συσκευέ στην αγορά και το ενεργειακό σήμα είναι σημαντικό. Το πρώτο λοιπόν, όποια ετικέτα τελικά αλλάξει, πρέπει να έχουμε μια αναθεώρηση και ένα σύστημα παρακολούθηση και αξιολόγηση μετά από τρία χρόνια. Για να δούμε αν αποδίδει. <clears throat> να δούμε αν κινεί την αγορά προς τα πιο αποτελεσματικά προϊόντα. Το πώς θα γίνει αυτό, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει για το περιβάλλον μεταφέρουν τι απόψει και των καταναλωτών και του Κοινοβουλίου ότι με αναθεώρηση A μέχρι G είναι ο πιο πρακτικός τρόπος για να είναι αποτελεσματικό το σήμα και όπως πολλοί είπανε αυτό πολλέ προηγούμενε εξολογήσει και έρευνε το επιβεβαιώνουν και μελέτη Γκάλεν και άλλε η έρευνα της Κομισιόν δείχνει κάτι διαφορετικό. Θα επανέλθω σε αυτό. Τονίζω ότι ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα ενό συστήματο A to G είναι ότι ένα προϊόν, αν είναι κακό, πρέπει να έχουμε σκληρή αξιολόγηση. Ένα σύστημα που επιτρέπει προϊόντα να φαίνονται σαν αλφα εντό εισαγωγικών και να δίνουν την εντύπωση στον κανητή ότι αγοράζουν κάτι που είναι φιλικό προς το περιβάλλον χωρίς να είναι. Αυτό είναι απάτη. Και είναι σημαντικό ρόλο που η μηχανία δεν θέλει αυτή την επιλογή. Τώρα, το αν θα οδηγήσει στο να κλείσουν εργοστάσια και να έχουμε πωλήσει όπω λένε οι βιομήχανοι, αυτό μέχρι στιγμή δεν το έχουν τεκμηριώσει. Τώρα έρχομαι στην έρευνα της Κομισιόν. Πρώτον, όπω ε, μα έδειξε η έκθεση του κ. Βεζέρη, η μεταβατική περίοδο μεταξύ των δύο ε, ετικετών παρουσιάζει δυσκολίε, Γιατί όποια από τι τρεις ετικέτες και αν επιλεγεί, το υλικό αποτέλεσμα ήταν λιγότερο από 50%. Ξέραμε ότι το πρόβλημα αυτό θα υπάρξει και μα παραξενεύει το ότι η Κομισιόν δεν φρόντισε να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Εμεί θέλουμε να συνεργαστούμε με όλου προκειμένου να βρεθεί λύση. Κανένα από τα σήματα αυτά βέβαια δεν είναι απόλυτα κατανοητό για την μεταβατική περίοδο. Το σύστημα κλώσ α έως g είναι αυτό που καταλαβαίνουμε λιγότερο. Αν ξαναδούμε τα slides, αν θυμηθούμε μάλλον τα slides που είδαμε πριν, ήταν πολύ μικρή η περίοδος και πολύ πιο μακριά το νούμερο αυτό από τα άλλα. Και στη συνάντηση που είχαμε και με την Κομισιόν για να συζητήσουμε πώς πρέπει να γίνει η έρευνα, ένα από τα feedback που είχαμε ότι η περίοδος αυτή επικύρωσης θα πρέπει να είναι στο κέντρο του σήματος με το γράμμα. Βέβαια αυτά τα σχόλιά μας δεν εγγύθησαν υπόψη. Επίσης η, με... η μεταβατική περίοδος πέρασε σε κατηγορία A, α, συν, συν. Φαίνεται λιγότερο καλό να περάσουμε από α, συν, συν σε α. Εν πάση περιπτώσει όμως, Το τεστ δεν ήταν και πάρα πάρα πολύ αντικειμενικό. Αυτά για την παρουσίαση του κυρίου Μπιζάν για τη μεταβατική περίοδο. Είναι κάπως μεροληπτική η παρουσίαση. Γιατί η μεταβατική περίοδος μεταξύ των σημάτων θα είναι μερικοί μήνες, αφού μιλάμε για τριετή περίοδο. Αν είναι λιγότερο από το 10% της ζωής του σήματος, αν και όπως είπε ο κύριος Φαρκιόνη, αν το δούμε αυτό στο σύνολο της αγοράς, σημαίνει ότι θα έχουμε συνεχώς μετάβαση γιατί δεν πάει ο καταναλωτή να αγοράσει όλα τα προϊόντα του με μιας. Και το πιο σημαντικό από τη μεταβατική περίοδο είναι από τη στιγμή που θα υπάρξει το σήμα πόσο κατανοητό θα είναι. Και αν δούμε το πρώτο σημείο της παρουσίας του κύριου Μπριζέρε. η δήλωση στα πορίσματα της παρουσίασης της Κομισιόν το Clause A μέχρι G είναι η πιο δυσνόητη κατά τη δική μας άποψη δεν στέκεται. Μία άλλη απόδειξη που χρησιμοποιήθηκε κατά του A του G είναι το πόσο δημοφιλές είναι. Και ρωτώ την Κομισιόν. Πώς ρωτήθηκε, πώς μπήκε η ερώτηση. Ήταν σαφές στον καταναλωτή ότι το ρωτήσατε όχι τι προϊόν προτιμούν, αλλά τι σήμα προτιμούν. η σύγκριση ήταν το α, είτε α συν συν, α μείον 40. Τι τους ρωτήθηκε. Όσο πιο λαμπρή φαίνεται η παρουσίαση στην ταξινόμηση, ε, τόσο λιγότερο γίνεται κατανοητή. Και έρχομαι στο τελική μου παρατήρηση όσον αφορά την έρευνα της Κομισιόν δεν είδε τους κύριους μάρτυρες. Είτε α συν είτε α 40. Οι ενδιαφερόμενοι είναι αυτοί που γνωρίζουν τα της αγοράς. Αν προσπαθήσω να αγοράσω ένα ψυγείο και έχει C σε ένα close I to G, ξέρω ότι θα πάω σε μια κατηγορία καλύτερα. είναι όμως α 40, πώς θα ξέρω αν θα κάνω καλύτερη επιλογή. Και όπως είπε η συνάδελφος από την BOIC, αν θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους καταναλωτέ να βράσουν τα καλύτερα προϊόντα, θα πρέπει το μήνυμα να είναι σαφέ. Και το buy α είναι σαφέ. Ενώ όμω πούμε ε, αγόρασε αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλε κατηγορίε, δεν είναι τόσο καθαρό αυτό το μήνυμα. Και ρωτήσαμε την Κομισιόν, βάλτε τέτοιες ερωτήσεις μέσα. Η Κομισιόν δεν το έκανε. Αυτά όσον αφορά την, ε, έκθεση, την έρευνα της Κομισιόν. Επαναλαμβάνω ότι χρειαζόμαστε μια επανεξιολόγηση οποιοδήποτε σχήματος επιλεγεί. Και το τελευταίο μου σχόλιο, σημαντικό όσον αφορά τι μη κυβερνικέ οργανώσει για το περιβάλλον, τα ε, μέτρα eco-design είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Χρειάζεται μεν το σήμα για να κατευθύνει τον καταναλωτή να αγοράσει καλά προϊόντα, αλλά τα μηνύματα eco-design αναφέρονται στο κατώτερο μέρος της αγοράς. Να απαλλαγούμε δηλαδή από τα χειρότερα προϊόντα. Δυστυχώς, μερικοί ισχυρίζονται ότι πρέπει αυτά τα δύο να αποφασίζονται παράλληλα για κάθε κατηγορία προϊόντων. Οι Κομισιόν και τα κράτη-μέλη αποφάσισαν να αναβάλουν και την ψήφο και για το eco-design μέχρι ότου επιληθεί το θέμα της ετικέτας του label που σημαίνει τα μέτρα eco-design για οι οικιακέ συσκευέ που είναι συσκευέ που καταναλώνουν πάρα πολύ ενέργεια θα περιμένουν το, τουλάχιστον μέχρι το Μάρτιο. Και όμως είναι σημαντικά για την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακος κλπ. Σας παρακαλούμε, λύστε το θέμα του της και συνεχίστε να δίνετε σημασία και στη διαδικασία για το eco-design. Τελειώνω με το εξή με τα εξή τρία. Πρώτον, για να καλυφθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι χρειαζόμαστε και καινοτομίε και επαναξιολόγηση και αναβάθμιση των προϊόντων που σημαίνει το ενεργειακό σήμα έχει σημαντικό ρόλο. Πρέπει το μήνυμα στον καντίνο είναι σαφέ για να αγοράζουν πιο αποδοτικά προϊόντα και να ξέρουν ποια είναι τα χειρότερα. Και αμφιβάλλουμε κατά πόσον ε, το open and scale μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Τουλάχιστον ε, δεδομένου ότι η έρευνα της Κομισιόν δεν, το, δεν έκανε αυτό τον έλεγχο. Και τέλος, όπως είπα, η κρίση ως να φρανιντικέτα δεν θα μπλοκάρει τη διαδικασία του eco-design. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και για την τοποθέτησή σας αυτή. Ακούσαμε τις διάφορες αξιολογήσεις και τα γεγονότα και τις γνώμες και μπορούμε να συζητήσουμε τα πράγματα μεταξύ μας λίγο. Υπάρχει δυνατότητα για συμπληρωματικές ερωτήσεις για δικές σας ε, τοποθετήσεις. Ε, θεωρώ το εξή σημαντικό. Ε, όλοι όσοι μίλησαν εδώ και έχει σημασία για το επόμενο διάστημα για μας ε, λέγουν ότι θα πρέπει να φροντίσουμε το συντομότερο δυνατό να περάσουμε στην εφαρμογή. Θέλουμε γρήγορα αποτελέσματα. Και ένα δεύτερο επίσης αδιαφυσβητητό ε, από το πάνελ αλλά και από την αίθουσα σίγουρα είναι ότι χρειαζόμαστε σήμανση, χρειαζόμαστε μια ετικέτα που να συμβάλλει και στην αποδοχή του κοινού και οι πολίτες να μπορούν γρήγορα να παίρνουν τη σωστή απόφαση και να αγοράζουν τις σωστές συσκευές. Γι' αυτά τα δύο συμφωνούμε. Η διαφορά μας πού είναι τώρα. Ποιο σήμα, ποια ετικέτα μπορεί να τα πετύχει αυτά. Ε, και διαφέρουν οι απόψεις και ακούσατε και τις έρευνες της αγοράς. Έχετε την ευκαιρία τώρα να μιλήσετε. Αν συμφωνείτε αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα στη Σουηδική Προεδρία στο βαθμό που θέλει να μιλήσει το Συμβούλιο και μετά εμείς. Καταρχήν επιθυμεί, όχι, δεν θέλει, δεν έχει να πει τίποτα η Σουηδική Προεδρία. Ωραία, πάει και αυτό. Πρόταση έκανα. Γιατί είμαι στον τριμερή διάλογο αυτό τον καιρό σχεδόν. Κοντεύει. Ωραία. Με τη σειρά που ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Μπριζίνα πρώτος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για ε, τη διοργάνωση αυτής της ακρόασης. Πολλά ε, καινούρια μάθαμε σήμερα. Για την κλίμακα αυτή για την ταξινόμηση θα ήθελα να σας πω ότι είπαμε μπορούμε να έχουμε μία ε, ανοιχτή ή κλειστή ε, κλίμακα. Η κλειστή ε, με τις κατηγορίες ε, α έως g ήταν καλή για αρχή όταν εισήχθη το σύστημα, όταν ξεκίνησε. Από όσα άκουσα σήμερα και από όσα κατάλαβα, εγώ θα προτιμούσα την ανοιχτή κλίμακα πλέον. Την α συν. Να σας πω και γιατί, ποια είναι τα επιχειρήματα. Τώρα δεν γνωρίζω πόσοι από εσάς... Ε, Αγοράσατε πρόσφατα οικιακή συσκευή με την νέα ετικέτα αυτή, γιατί κυκλοφορεί στην αγορά. Είχα πάει λοιπόν σε ένα κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και έχω προσωπική εμπειρία. Σχεδόν όλοι οι κατασκευαστές πλέον παράγουν συσκευές που έχουν χαρακτηρισμό α, ε, τουλάχιστον αυτές που κυκλοφορούν στα καταστήματα. Και η μόνη δυνατότητα ε, να διαπιστώσει κανείς διαφορά ήταν η ανοιχτή κλίμακα προς τα πάνω. Ε, ο κύριος Φαντσόν μίλησε για τα νέα προϊόντα στην τελευταία έκθεση του Αμβούργου και ακριβώς είναι πιο οικολογικό αυτό το σήμα, θεωρώ εγώ. Στη συνέχεια ακούσαμε και για τους ε, πολιτές που μιλούν στους καταναλωτές και τους ενημερώνουν για το α μείον ε, χ της 100 και όντως μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Όταν όμως είναι κλειστή η κλίμακα, λες, ε, αυτή η συσκευή είναι κατηγορίας α. Ναι, κατηγορίας α όταν παρήχθη. Τι γίνεται όμως με τα νέα προϊόντα που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά. Αυτά είναι α-50, δεν υπάρχει α. Καλύτερο λοιπόν να έχουμε τη, τη δεύτερη κατηγορία με το συν, α συν ή α συν συν, για να καταλαβαίνει ο καθένας πιο εύκολα και να αποφασίζει πιο εύκολα. Και το χρώμα, το πράσινο επίσης είναι μεγάλο κίνητρο. Οικολογικοί λοιπόν πρωταθλητές ε, από πλευρά των συσκευών θα έχουν καλύτερη σήμανση. Μου προκαλεί έκπληξη το γεγονό ότι οι πράσινοι οικολόγοι και οι πράσινες κατά τα άλλα μη κυβερνητικέ οργανώσεις δεν επιλέγουν αυτή την ανοιχτή κλίμακα. Την η Είναι και πιο οικολογική και πιο κατανοητή και εύληπτη για τους καταναλωτές. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα λοιπόν εμείς θα προτείνουμε να υποστηριχθεί η ανοιχτή αυτή κλίμακα οπωσδήποτε Ευχαριστώ. Ε, η κυρία Χολ παρακαλώ. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχω απογοητευτεί εγώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έρευνά της. Και βαθιά. Διότι θεωρώ ότι έγινε μια απόπειρα εδώ να χειραγωγηθεί η πολιτική απόφαση. Η πολιτική απόφαση των Ευρωβουλευτών ήταν σαφής. Το βασικό ερώτημα ήταν το εξής. Θέλουμε κλειστή κλίμακα με αναθεώρηση ναι ή ου. Και οι βουλευτές αποφάσισαν ότι θέλουν κλειστή κλίμακα. Θέλουμε κλειστή κλίμακα γιατί τελικά το ζήτημα ποιο είναι. Θέλουμε ο κόσμος να ξέρει ότι είναι σχετικό το να είναι ένα προϊόν καλό για το περιβάλλον. Κάτι που είναι καλό σήμερα μπορεί μετά από πέντε χρόνια να μην είναι πια καλό σε σύγκριση και σχέση με νέα προϊόντα. Αν δεχθούμε ότι είναι σχετικό αυτό το καλό ή το κακό για το περιβάλλον και αλλάζει, τότε θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αναθεωρείται η κατάταξη αυτή αυτό δεν το δέχεται η βιομηχανία. Και τι έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έρευνα. Τα έκανε πλακάκια με τη βιομηχανία ακολούθησε αυτή τη τακτική ότι δεν θέλουν αναθεώρηση της κλίμακας και αγνόησε τους εκλεγμένους βουλευτές που είπαν ότι θέλουν κλειστή κλίμακα με αναθεώρηση για να ε, αποκομίζουμε τα περισσότερα ωφέλη όσο γίνεται από την ετικέτα. Λοιπόν, εγώ έχω το εξή βασικό πρόβλημα ε, με την έρευνα. Κάνετε λάθος ερωτήσεις. Θα μπορούσατε να έχετε ερωτήσει πολλά πράγματα για την αναθεώρηση της κλίμακας με επιλογές, ας πούμε ημερομηνίε, ε, με μεγαλύτερη προθεσμία ή να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση ε, στην κατανάλωση για να γράφει η ετικέτα την κατανάλωση και να συγκρίνουν οι καταναλωτές δύο ετικέτες που να λένε ότι είναι β για παράδειγμα αλλά πουθενά δεν ανάγεται η διαφορά, δεν γράφεται η διαφορά στην κατανάλωση. Θα μπορούσαν πολλά στοιχεία να δοθούν στους καταναλωτές για να αποφασίσουν, για να απαντήσουν και δεν τους δόθηκαν. Επίσης πιστεύω κάτι ακόμα, ότι μας προκαλεί έκπληξη. Μπορεί και να μην μας προκαλεί βέβαια, ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας. Πάντως υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα ε, στις, ε, στα ευρήματα αυτών, αυτής της έρευνας με εθνικές έρευνες που με τρόπο πιο ευθύ προσπάθησαν στα κράτη-μέλη να βρουν ποιος είναι ο πιο εύκολος ε, τρόπος να καταλαβαίνουν οι καταναλωτές. Εδώ υπάρχει μια ερώτηση που γίνεται μόνο στους καταναλωτές που κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται. Όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν που δεν κατάλαβαν το μοντέλο δεν απαντούν στην επόμενη ερώτηση. Μα τι στο καλό έρευνα είναι αυτή. Εμείς ως πολιτικοί θα ε, καταλαβαίνουμε όλα αυτά πολύ καλά γιατί Ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά ο κόσμο θέλει απλά πράγματα, να το εξηγεί. Αυτό το ευρωπαϊκό σήμα είναι και παγκόσμια προδιαγραφή και είναι πολύ απαραίτητο, όχι μόνο για την ευρωπαϊκή εξονόμηση ενέργεια, αλλά ε, και παγκοσμίω. Και είναι πολύ απλό το σήμα, γιατί κινδυνεύουμε τώρα το εξή. Να χάσουμε όλα τα πλεονεκτήματα που μπορούμε να έχουμε, που βάζουμε και συγκριτική αξιολόγηση και benchmark, αν τα θαλασσώσουμε εδώ. Πραγματικά σας λέω ότι έχω απογοητευτεί βαθύτατα που έγινε με αυτόν τον τρόπο η έρευνα. Και δεν ελήφθη υπόψη η βασική πολιτική απόφαση που είχε ληφθεί εδώ στο Κοινοβούλιο. ευχαριστώ. Ο σύναφος Σόζα Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω ε, τις παρουσιάσεις που έκαναν ε, σήμερα μιλητές μας ήταν πολύ λεπτομερείς και εύστοχες και μου επέτρεψαν και μένα να μάθω τα, ε, το ιστορικό του θέματος αυτού. Σε δεύτερο λόγο θέλω να ζητήσω συγγνώμη και από τους ηγητές και από τους υπολείπους συναδέλφους βουλευτές γιατί θα κάνω μια ερώτηση αρκετά απλή. Αλλά είμαι και νέο μέλος στο Κοινοβούλιο και δεν γνωρίζω πάρα πολύ καλά το ιστορικό όπως σας είπα και τι προηγήθηκε. Θα ήθελα να μάθω συγκεκριμένα στο σχέδιο οδηγίας τι χώρο έχουν, τι ελευθερία κινήσεων έχουν να δράσουν τα κράτη-μέλη για να ρυθμίζουν αυτό το θέμα. Θα ήθελα να το γνωρίζω αυτό και να σας πω και γιατί. Όσο λιγότερη ελευθερία έχουν τα κράτη-μέλη, τόσο το καλύτερο. Αλλά θα ήθελα να μάθω τι ε, λέει αυτό το σχέδιο. Τα κράτη-μέλη τι ευκαιρία έχουν. Μπορούν να μου το εξηγήσουν αυτό πολύ σύντομα παρακαλώ και πολύ απλά. Ναι, θα ήθελα να απαντήσω. Ο λόγος που γίνεται όλη αυτή η άσκηση είναι να υπάρχει μία ενιαία ρύθμιση σε όλη την Ευρώπη. Ο κύριος Λάγκερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να ρωτήσουμε γιατί γιατί επισημούμε η Κομισιόν επισημεί μια ανοιχτή κλίμακα. Για μένα ο μόνος λόγος πίσω από αυτό είναι ότι η βιομηχανία, ο βιομηχανικός τομέας θέλει να αποφύγει ε, την ε, σήμαση των προϊόντων με κόκκινο. Σήμερα ακούσαμε τι ωραία που είναι όλα τα πράγματα με την πράσινη ετικετοποίηση, πράσινη κλίμακα. Εάν λοιπόν γράψουμε στα προϊόντα αυτά την καινούργια ετικετοποίηση 50, ε, 60, οτιδήποτε όλα τα προϊόντα θα βγουν πράσινα, ωραία και καλά. Άρα δεν παρουσιάζουμε καμία ε, ε, σωστή επιλογή για τον καταναλωτή εγώ προτιμώ μία κλειστή κλίμακα η οποία θα έχει πράσινο, κίτρινο κόκκινο και αυτή είναι μια διαφανής και ειλικρινής μέθοδος. Δεν πιστεύω ότι ένας καταναλωτής, αν τον ρωτήσουμε ποια ετικέτα επισημεί, Ε, και άμα του πούμε ταυτόχρονα ότι όλε, όλες οι ταξινομήσεις είναι πράσινες έτσι κι αλλιώς και ποια επιθυμεί από αυτές τις πράσινες δεν έχει και νόημα, είναι άνευ αυτή η επιλογή. Γι' αυτό θέλουμε κλειστή ταξινόμηση, κλειστές κλίμακες διότι με το σύστημα της κλειστής ταξινόμησης θα μπορέσουμε να προβάλλουμε τη βιομηχανία εκείνη η οποία πραγματικά παρουσιάζει και κατασκευάζει τις καλύτερες συσκευές. Η κυρία Ρία Ραμαντουρέλ, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και εγώ πολύ σύντομα θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους ομιλητές μας για την παρουσία και τις παρουσιάσεις τους. Και όλο ιδιαίτερο στην κυρία Ποδηματά θα ήθελα να συγχαρώ για τη καλή δουλειά που κάνει σε αυτό το θέμα τόσο καιρό για ε, τις ετικέτες. Είναι πολύ σημαντικό για την εξοικονόμηση ενέργειας αυτό. Θέλω επίσης να σας πω ότι μας βοηθάει πάρα πολύ για τη δουλειά μας και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσουμε τι λένε οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς και οι διάφοροι κλάδοι. Για τη δική μας πολιτική ομάδα είναι επίσης πολύ σημαντικό να έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και τις οργανώσεις των καταναλωτών. Έτσι ώστε να μπορούμε να πάρουμε τις αποφάσεις μας με τα λόγου γνώσεως και να ξέρουμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες. Ευχαριστώ και πάλι ε, τους εκπροσώπους των καταναλωτικών οργανώσεων για τις ε, απόψεις σας. Εγώ θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις και κάποια σχόλια πάρα πολύ απλά. Με όλες τις επιφυλάξεις που εξέφρασε η κυρία Χορ, εμένα μου φάνηκε πολύ χρήσιμη η διευκρίνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πώς έχει κατάσταση και τι γίνεται, πώς καταλαβαίνει ο κόσμος τις ετικέτες. Για να βελτιωθεί όμως ακόμα πιο γρήγορα η κατανόηση θα βοηθούσε πάρα πολύ να είμαστε κατηγορηματικοί και να παρέμβουμε στα σχολεία, στην παιδεία αλλά και στη διαβίου εκπαίδευση. Να ενημερώνει το καταναλωτής. Γιατί επανειλημμένα ακούμε στη συζήτηση και βλέπουμε να εμφανίζεται ε, η μορφή του πολιτή. Ο πολιτής που έρχεται να διαγωγήσει και να εκπαιδεύσει τον καταναλωτή. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο ο πολιτής. Μπορεί να τους δώσει ε, στοιχεία, εξηγήσει Βεβαίω και υπάρχει ετικέτα ανάμεσα στον κατασκευαστή και στον αγοραστή, αλλά υπάρχει και ένα πρόσωπο ενδιάμεσο που λέγεται πολιτή και έχει κατάρτιση, εκπαίδευση και είναι η δουλειά του. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω και οι κατασκευαστέ και οι καταναλωτέ τι έχουν κάνει, έχουν ε, αναλάβει καμιά πρωτοβουλία για να εκπαιδεύουν το προσωπικό τους πολιτές των συσκευών αυτών που είναι σε επαφή με το κοινό. Άλλη ερώτηση και πάλι ε, την απευθύνω και στους κατασκευαστέ, και στου καταναλωτέ. Από ό,τι φαίνεται είναι προφανής και αυτονόητο και το έχω κατάλαβει και εγώ ότι χρειάζεται αναθεώρηση, ανανέωση η ετικέτα και τακτική. Ε, οι κατασκευαστές ρωτάνε ποιος φέρει την ευθύνη αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί ε, στα μαγαζιά και στο εμπόριο η συσκευή. Αλλά εγώ θα ήθελα να μάθω το πραγματικό κόστος ενημέρωσης κάθε φορά της ετικέτας. Ή η σχέση κόστος-οφέλους αν θέλετε. Γιατί έχω αντιφατικές ε, πληροφορίες και ενημέρωση και θα ήθελα να μάθω τι λένε οι κατασκευαστές και οι καταναλωτές γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ. Ο κύριος Τσίτσεστερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την κυρία Ποδηματά που οργάνωσε αυτή την ακρόση. Και ευχαριστώ και όλους τους ομιλητές για τις εισηγήσεις τους. Ομολογώ ότι ε, έχω μια επιφύλαξη προσωπική για την προσέγγιση αυτή η οποία μοιάζει με τα σήματα, τα φανάρια της τροχέας. Ε, είναι λίγο απλοϊκή, αλλά δεν θα το αναπτύξω σε βάθος. Η κλειστή λίστα, η κλειστή κλίμακα, εάν επαναξιολογηθεί πιστεύω ότι θα οδηγήσει σε καταχρήσεις και μεγάλη σύγχυση, μεγάλο μπέρδεμα όταν θα θέλουμε να πληροφορήσουμε σωστά και εύκολα τους καταναλωτές μας. Η, σημείωσα ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις είναι επιφυλακτικές ως προς τις μελέτες της Κομισιόν. Ξέρουμε τώρα ότι οι σφιγμομετρήσεις και ε, τα ερωτηματολόγια είναι κατευθυνόμενα από τις ερωτήσεις που περιέχουν και πολλές φορές οδηγούν προς μία κατεύθυνση μέσω των απαντήσεων. Άρα λοιπόν ε, κάθε φορέας που παρουσιάζει ένα τέτοιο ερωτηματολόγιο μπορεί να είναι λίγο ύποπτος. Αυτή τη στιγμή όμως η απάντηση της Κομισιόν δεν είναι, δεν μας βοηθάει. Δεν μας βοηθάει ιδιαίτερα ε, σε σχέση με την αρχική της πρόταση, το α μείον, ε, Δεν είναι σαφές αυτό το α ε, τι είναι ακριβώς και πιστεύω ότι μπορεί να είναι παραπλανητικό. Γι' αυτό εγώ, και δεν θα σας εκπλήττει, προτιμώ το α συν συν. Πιστεύω ότι το α με ένα διπλό συν είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τη μεταβατική περίοδο με τη νέα αξιολόγηση. Είναι, είναι δύσκολο θέμα. Ε, δεν νομίζω να υπάρχει απλή λύση και σαφώς συμφωνώ με την κυρία Χαουπ. Πρέπει να καταλήξουμε σε μία απόφαση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Γιατί συμφωνώ με τους συναδέλφους που είπαν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προβάλλουμε και να ενισχύσουμε την ε, ενεργειακή απόδοση, μια καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Και μια τελική παρατήρηση. Την τελευταία φορά που αγόρασα μια συσκευή, είχα δύο πράγματα υπόψη μου. Ε, το πρώτο είναι να προσέξω την ενεργειακή ταυτότητα και το δεύτερο βεβαίως κριτήριο ήταν το κόστος. Ασφαλώς ε, θέλω να έχω την καλύτερη ενεργειακή απόδοση αλλά και την καλύτερη τιμή. Ε, υπάρχει, υπάρχουν λοιπόν διάφορες ε, απόψεις των καταναλωτών και διάφορα κριτήρια κυμαίνονται τα κριτήρια των καταναλωτών. Εγώ εμένω στην υιοθέτηση της μεθόδου α συν συν αυτής της κλίμακας. Ευχαριστώ. Κύριο Ζαντό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μερικές παρατηρήσεις. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η μέθοδος της Κομισιόν εστιάζεται κυρίως στην κλειστή λίστα όσο και στην περίοδο τη μεταβατική. Ίσως καταλαβαίνουμε υπερβολικά καλά ότι πρόκειται για μια προσπάθεια να δοθεί μια απάντηση διασφάλισης για τους βιομήχανους παρά να φτάσουμε στον στόχο αυτής της διαδικασίας, δηλαδή να δώσουμε αναγνωσιμότητα, ορατότητα και απλοποίηση στην αναγνώριση εκ μέρους των καταναλωτών της ετικέτας. Γιατί καλό είναι οι ετικέτες να είναι κατανοητές αυτό θα επαναπροσανατολίσει τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Των καταναλωτών. Πρώτη ερώτηση λοιπόν προς την Κομισιόν. Γιατί εστιάζετε τόσο πολύ στη μεταβατική περίοδο και επικρίνατε τόσο πολύ την κλειστή ε, ταξινόμηση με βάση μόνο αυτό. Δεύτερο, ερώτηση προς την Κομισιόν πάλι. Η ανάλυση για τα μειονεκτήματα της ε, ανοιχτής ταξινόμησης. Δεν το πολύ καταλαβαίνουμε. Βλέπουμε τους κινδύνους. Έχω εδώ μία διαφήμιση της Electrolux που παίζει πολύ με την ανοιχτή, ποντάρει πολύ στην ανοιχτή ταξινόμηση. Να σας δώσω τα πρώτα πέντε αποτελέσματα στην αφάντη την κατηγορία. ρούχων. Α πλούς Α'. Το δεύτερο άνα Α πλούς πλούς Α'. Τρίτο Α συν συν ΑΜΠ. Τρίτο Α και το πέμπτο ΑΑΑ αυτά. Εμείς θεωρούμε την εσωτερική λογική της ανοιχτής ταξινόμησης. Δηλαδή, ο κατανοητής χάνεται εντελώς μέσα σε όλα αυτά τα γράμματα και νούμερα. Άλλη ερώτηση προς την Κομισιόν. Στην παρουσίασή σας μας λέτε πάνω από το 70% του δείγματός σας θεωρεί ότι η κλειστή ταξινόμηση είναι ενδιαφέρουσα. Στα πορίσματα μας όμως θεωρείται ότι αυτό παρουσιάζει μειονεκτήματα. Πώς περνάτε, με ποια λογική ακολουθία περνάτε από την πρώτη σκέψη στη δεύτερη. Κάτι άλλο. Αναφέρθηκε ότι ζητήθηκε γνώμη των ενώσεων και ότι έγινε με διαβούλευση. Πείτε μας κάτι παραπάνω. Έγινε αυτή η διαβούλευση. Πώς έγινε. Και πώς οι παρατηρήσεις σας ε, εμπλουτίστηκαν από αυτό και αν ελήφθησαν υπόψη. Αυτή τη στιγμή συζητάμε το θέμα ετικέτες για τα ελαστικά αυτοκινήτων και νομίζω εκεί για η Κομισιόν υιοθέτησε κλειστή ταξινόμηση. Πώς συμβιβάζεται αυτό με τη θέση που παίρνει εδώ η Κομισιόν όσον αφορά την ετικέτα. Και τέλος, εμείς κάναμε και εμείς μια έρευνα δική μας στο Ευρωκοινοβούλιο με ερώτημα τι είναι πιο εύκολο, τι είναι πιο χρήσιμο. 54% ήταν κλειστή λίστα ΑΖ. Αυτές οι παρατηρήσεις μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ο κύριος Καντσιάν. Ελπίζω να το είπα σωστά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για όλη την προσπάθεια η οποία καταβλήθηκε. Εγώ πρώτη φορά ακούω σχετικά με το θέμα αυτό και θεωρώ ότι ορισμένε σκέψεις είναι σκόπιμα να γίνουν. Βλέπω ότι υπήρξε έντονη δέσμευση προκειμένου να επιτευχθεί ένας στόχος εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό ήταν ο κύριος στόχος. Έχω την εντύπωση ότι φορτώνουμε στους καταναλωτές κάτι που έπρεπε να λυθεί πιο πριν, πιο νωρίς, όχι στο επίπεδο του καταναλωτή. Αναφέρθηκαν προβλήματα που αφορούν την περίοδο μεταξύ παραγωγής και χρήσης του προϊόντος Παραμένει όμως μια αμφιβολία ως προς αυτό. Έπειτα η επικαιροποίηση στις διάφορες ετικέτες. Εγώ πιστεύω ότι αν λάβουμε υπόψη το στόχο που είναι η εξοικονόμηση θα πρέπει να προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα εγκαίρως απλοποιώντας τα πράγματα, δηλαδή να δείξουμε λίγο παραπάνω θάρρος και για αυτούς που παράγουν και για αυτούς που πουλάνε τα προϊόντα. Μην βάλουμε τον κατανοητή σε μια κατάσταση που να μην μπορεί να καταλάβει ή να πάει να επιλέξει κάτι που, που δεν είναι απλό για αυτόν. Δηλαδή, πρέπει να προσπαθήσουμε οι ετικέτες αυτές είναι προσανατολισμένες προς την αποδοτική χρήση της ενέργειας και προς ένα πιο απλό μοντέλο. Από τα τρία μοντέλα που ελέγχθηκαν βλέπω ότι το κλειστό μοντέλο έχει 13% των καταναλωτών, το ΑΣΥΝ 40% και το τρίτο 43%. Βλέπουμε δηλαδή ότι εδώ υπάρχει μια αντίφαση στην απάντηση των ίδιων των καταναλωτών στην κλειστή ετικέτα ε, το ποσοστό είναι μικρότερο, το ποσοστό υπέρ. Εγώ αυτά τα στοιχεία δεν μπορώ να τα συμφιλιώσω, δεν το καταφέρνω. Γιατί πιστεύω ότι όποιος πάει να αγοράσει ένα τέτοιο προϊόν πρέπει να έχει μπροστά του κάτι πολύ πιο απλό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, δυστυχώς παρέβλεψα τον αντιπρόεδρό μας, τον κύριο Ρόντε. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω ε, στα δανέζικα και παρακαλώ χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σας, αν θέλετε να με ακούσετε. Έχω ε, δουλέψει μερικά χρόνια στο διαφημιστικό τομέα και ε, είναι σαφές. Εάν θέλουμε να πουλήσουμε περισσότερα πράγματα, αν θέλουμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά των καταναλωτών, πρέπει οπωσδήποτε να ακούσουμε τη φωνή των καταναλωτών. Και λύσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη αυτή τη φωνή των καταναλωτών δεν αξίζουν, δεν έχουν καμία αξία. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να ακούσουμε τους καταναλωτές εδώ. Έχει αποφασιστική σημασία και επίσης να παρουσιάσουμε ένα προϊόν όσο το δυνατόν πιο απλά. Η η απλότητα, η, εύκολη κατανόηση είναι το πρώτο βήμα. Και εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι πρέπει να παραμείνουμε σε ένα κλειστό σύστημα για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την απλότητα. Ιδίω τώρα που άκουσα πώς ένα ανοιχτό σύστημα θα δημιουργήσει σύγχυση, ε, τότε παρουσιάζεται ο κίνδυνος οι καταναλωτές να συμπεριφερθούν πολύ διαφορετικά από ό,τι εμείς ε, επισημούμε. Τώρα η ερώτηση είναι πρέπει να περιπλέξουμε τα πράγματα τόσο πολύ, δεν μπορούμε να βρούμε έναν απλούστερο τρόπο. Μία ετικέτα με μία χρονολογία. Και από πλευράς κομισιών θα πρέπει μαζί με τον βιομηχανικό τομέα, με τον ενδιαφερόμενο τομέα, να καθορίσουμε μία προθεσμία, μία, ένα έτος όπου μέχρι τότε να μπορέσουμε βαθμιαία να καταλήξουμε στο τι πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε τελικά σε ένα αποκλειστικά πράσινο περιβάλλον. Δηλαδή βαθμιαία, χρόνο με το χρόνο, σιγά σιγά να βλέπουμε μέχρι μια χήμερομηνία, πότε θα καταλήξουμε σε ένα απόλυτα πράσινο περιβάλλον. Έτσι ώστε και ο καταναλωτής να καταλαβαίνει τα πράγματα και τις κλίμακες. Ωραία, μπορεί ίσως η, ο τομέας της ε, βιομηχανίας να μην του αρέσει πολύ αυτή η λύση, αλλά ε, δικός μας στόχος είναι η Πλούστευση, η διαφάνεια, η εύκολη κατανόηση των καταναλωτών, διότι μόνο έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε την πώληση συσκευών που έχουν την καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Του τεστ είναι ο στόχος μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Τίκαου έχει την, τον τελευταίο λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς την κυρία Ποδηματά για την ε, εισήγησή της και για την πρωτοβουλία της να διοργανώσει αυτή την ε, ακρόση στην Επιτροπή μας. Υπάρχουν ολισμένα κράτη, και δεν μιλώ μόνο για κράτη-μέλη της Ένωσης, που για να προωθήσουν τις ε, πωλήσει συσκευών προσφέρουν επιδοτήσεις επιδοτούν δηλαδή την ε, πώληση προϊόντων, κατασκευή και πώληση. Επιδοτούν μάλιστα συσκευές ε, της ε, χειρότερης απόδοσης, της ενεργειακής απόδοσης, δηλαδή της χειρότερης ποιότητας συσκευές. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει οι ετικέτες και η ενεργειακή ταυτότητα να είναι όσο το δυνατό πιο εύκολα κατανοητή και απλή. Γιατί ένας καταναλωτής ε, θα αγοράσει ένα καλύτερα ενεργειακό προϊόν. Γιατί, διότι ξέρει ότι θα ξοδέψει λιγότερη ενέργεια, θα προστατέψει το περιβάλλον και θα πληρώσει και λιγότερο λογαριασμό. Ε, εγώ υποστηρίζω την πρόταση της κυρίας εισηγήτριας και πιστεύω οι διαβουλεύσεις που θα γίνουν με το Συμβούλιο θα καταλήξουν σε μια σωστή οδηγία η οποία θα ωφελήσει τους καταναλωτές. Διότι εάν τελικά υιοθετηθεί ένα περίπλοκο σύστημα με υπερβολικές πληροφορίες το οποίο δεν είναι σαφές, είναι συγκεχημένο, δεν ακολουθεί ξεκάθαρα κριτήρια, τι θα επιτύχουμε, το να μπερδευτούν τελείως οι καταναλωτές και το να προδώσουμε τους ε, στόχους μας για την ε, βέλτιστη ενεργειακή απόδοση. Εγώ πιστεύω ότι η έκθεση της κυρίας Ποδηματά συνδέεται άμεσα και με την ενεργειακή απόδοση κτηρίων. Το σώμα μας έχει ζήτησε και πέτυχε στην οδηγία αυτή να περιληφθούν minimum standards, minimum πρότυπα και προδιαγραφές για τα οικοδομικά υλικά έτσι ώστε να υπάρξει βέλτιστη ενεργειακή απόδοση στα κτίρια. Μπορούμε το ίδιο να το κάνουμε και για αυτή την οδηγία για τις συσκευέ. Ευχαριστώ. Μα γι' αυτό ακριβώς κάναμε ακρόαση σήμερα για να ακούσουμε τα ευρήματα των νέων ερευνών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τα αξιολογήσουμε και να δούμε. Προσπαθήσαμε να δούμε τι κάνουν οι καταναλωτές και πώ βλέπουν τη νέα ε, κατάταξη. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, όχι πάρα πολύ και θα παρακαλούσα τώρα όλου του ομιλητέ του πάνελ είτε να απαντήσουν σε ερωτήσει είτε να τοποθετηθούν γιατί έγιναν και κάποια ερωτήματα. Αν συμφωνείτε να αρχίσουμε τώρα εξ αριστερών προ τα δεξιά. Η κυρία Χόπ είναι πρώτη. Η Χόουπ, πώ σα λένε, ακόμα δεν έμαθα. Χόουπ, είναι το σωστό. ωραία. Η σειρά σα τώρα. Συγγνώμη που πρέπει να το μάθω το όνομά σα, δεν το έχω χωνέψει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα τα σχόλιά μου για τον κύριο Μπρεζίνα σχετικά με το θα έχουμε νέα προϊόντα στην κλίμακα. Κάθε φορά από το ASG το σχήμα θα ξαναορίζεται να υπάρχει χώρο στην άνω μέρος να μπουν νέα προϊόντα. Ένα νέο προϊόν φαντάζομαι θα είναι καλύτερο αν ήταν α και αν άλλο προϊόντα φαίνεται χειρότερα B, C, D παρά αν όλα προς τα κάτω ήταν α ή α συν ή α συν συν. Για την κυρία Χολ, συμφωνώ με όλα τα σχόλιά σας. Δυστυχώς θεωρούμε ότι η έρευνα της Κομισιόν δεν αποτελεί πλήρη βάση για απόφαση. Πολλές σημαντικές ερωτήσεις δεν ετέθησαν η επίπτωση στην επιλογή μεταξύ διαφόρων προϊόντων, που αυτό υποτίθεται ότι είναι στόχο τη ετικέτα. Για τον κύριο Λάγκε, συμφωνούμε απόλυτα ότι το πράσινο χάνει το νόημά του αν όλα έχουν α στον τίτλο. Ένα καλό τεστ θα ήταν πόσο μπορούμε να πάμε όσον αφορά την κορυφή στην κλίμακα. Για την κυρία Ριέρα Μαντουρέλ, συμφωνούμε ότι οι κατασκευαστές και οι πολιτές πρέπει να εκπαιδευτούν αλλά και οι καταναλωτές πρέπει να καταλαβαίνουν την ετικέτα buy α είναι ένα απλό μήνυμα για τον καταναλωτή όσον αφορά το κόστος θα πρέπει να διερωτηθούμε ποιο θα είναι το κόστος αν δεν προωθήσουμε τέτοιες συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας για τον κύριο Τσίτσεστερ αν λάβουμε υπόψη ότι το κόστος λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να αγοράσει κάποιος μια συσκευή εξοικονόμησης ενέργειας τονίζονται τα κακά προϊόντα και δεν είδαμε από την Κομισιόν μια κίνηση αντίστοιχη. Δηλαδή, με δύο λόγια, δεν πρέπει τα κακά προϊόντα να φαίνονται ότι είναι καλά. Για τον κύριο Ζαντό, για τη διαβούλευση της Κομισιόν, σας ευχαριστούμε που το δηλώσετε αυτό, διότι είμαστε απογοητευμένοι. Οι εκπρόσωποι μας πήγανε στη συνάντηση αυτή η διαβούλευση κάναμε σχόλια για την ανάγκη ερωτήσεων για τα προϊόντα στην κορυφή της πυραμίδας δεν ελήφθησαν υπόψη ούτε καν δεν μας έστειλαν τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας άρα ήταν κάπως μικρόψυχη αυτή η διαβούλευση για τον Ισπανό ή Ιταλό δεν ξέρω ευρωβουλευτή αν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα πιο έγκαιρα όπως και για το eco-design και για τον κύριο Ρόντε, τον αντιπρόεδρο, συμφωνούμε απόλυτα ότι οι καταναλωτές, οι καταναλωτές θα καταλάβουν το θέμα της μεταβατικής περίοδου και είναι κρίμα το ότι αυτό αναφέρεται με πάρα πάρα πολύ μικρά γράμματα. Με άλλα λόγια υπήρξαν πολλές επιλογές που δεν ελήφθησαν υπόψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επειδή ο κύριος Τζόνς πρέπει να φύγει, θα δώσω το λόγο σε εκείνον εκ μέρους της Κομισιόν, επειδή υπήρχαν πολλές ερωτήσεις που το απευθύνθηκαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για όλα τα σχόλια και τις ερωτήσεις. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμα λάβει απόφαση. Μα ζήτησαν να συντάξουμε μία μελέτη, να κάνουμε μία διαβούλευση και να συζητήσουμε το θέμα πρέπει να πω ότι υπογοητεύτηκα λίγο, στεναχωρήθηκα λίγο με τα σχόλια της κυρίας Χόουλ. Κάναμε μία ειλικρινή προσπάθεια να απαντήσουμε σε δύο ερωτήματα. Πρώτον, ποιες από τις διαφορετικές ταυτότητες τις καταλαβαίνει καλύτερα ο καταναλωτής έχοντας υπόψη τις πληροφορίες που θέλουμε να του μεταδώσουμε. Και δεύτερον, Τι καταλαβαίνει ο καταναλωτής ε, όταν, θα όταν μετακινούμαστε από το, από το ένα σύστημα στο, άλλο. Θα καταλάβει καλύτερα το, το σύστημα α προς β ή το α προς α συν συν. Αυτό το οποίο δεν κάναμε είναι να θέσουμε ερωτήσεις οι οποίες θα μας έδωναν απαντήσεις τέτοιες ώστε να κατευθύνουν τον καταναλωτή προς την α ή β απάντηση. Δεν προσπαθήσαμε να χειραγωγήσουμε τους καταναλωτές της απαντήσεις σας και ορισμένες από τις ερωτήσεις που οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις μας ζήτησε να συμπεριλάβουμε στα ερωτηματολόγια και στις φυγομετρήσεις έλεγαν ή έδειχναν μάλλον προς μία κατεύθυνση. Δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να, να πείσουμε τον καταναλωτή να απαντήσει προς την μία ή την άλλη κατεύθυνση παρά να τον αφήσουμε να έχει μία ελεύθερη επιλογή. Κατευθυνόμενες δηλαδή ερωτήσεις. Ενώ εμείς αυτό που θέλουμε να καταλάβουμε είναι ποιος τύπος ενεργειακής ταυτότητας ετικέτας είναι πιο εύκολα κατανοητή το α ή το ή β, ποια κατηγορία, ή το α συν συν. Η Κομισιόν πιστεύουμε ότι αυτό είναι ο στόχος ε, της ε, ταυτότητας, η εύκολη και ειλικρινής κατανόηση και όχι η χειραγώγηση του καταναλωτή. Αυτά είχα να πω ε, εισαγωγικά. Τώρα, ο Επίτροπος και η Εκτελεστική Επιτροπή δεν έχουν λάβει καμία απόφαση μέχρι τώρα και είμαι λίγαν απογοητευμένος όταν μου λέτε ότι η Κομισιόν προσπαθεί μεροληπτή μάλλον προς μια κατεύθυνση και σπρώχνει ε, όλη την υπόθεση προς την μία κατεύθυνση. Το αρνούμε αυτό. Εμείς θέλουμε να καταλήξουμε στην, στο καλύτερο, στον καλύτερο τρόπο για να δίνει ο καταναλωτής μία ενημερωμένη, πληροφορημένη και ε, σωστή απάντηση, να έχει μία σωστή επιλογή. Η ερώτηση είναι, οι πληροφορίες που περιέχονται μέσα στην ετικέτα παρέχουν ε, στον καταναλωτή τη δυνατότητα να λάβει μία σωστή ε, απόφαση. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και όχι να χειραγωγήσουμε και να κατευθύνουμε τον καταναλωτή να αγοράσει το α ή το β. Όχι, θέλουμε να πάρει μία intelligent decision, μία έξυπνη απόφαση. Και με τον τρόπο αυτό τον, της προτίμησης των καταναλωτών να ε, δείξουμε το δρόμο στην ε, βιομηχανία να παράγει καλύτερες συσκευές και πιο αποδοτικές. Προσφορά και ζήτηση δηλαδή. Πιστεύω ότι η μελέτη της Κομισιόν παρουσιάζει πάρα πολλά πληροφοριακά στοιχεία. Δεν λέμε ότι είναι το α και το ω όλων των, η βίβλος όλων των ε, μελετών. Όχι. Ε, εξετάσαμε σωρία άλλων μελετών και ερευνών που υπάρχουν στη διάθεσή μας για να παρουσιάσουμε την πρότασή μας στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Ε, εμπεριστατωμένη μελέτη κάναμε για να συντάξουν αυτή την ε, έρευνα. Δεν ξέρω, Άντρε, θέλει να προσθέσει. Να απαντήσω σε μερικά ερωτήματα που ετέθησαν στην Κομισιόν. Πρώτον, γιατί εστιαζόμαστε τόσο πολύ στη μεταβατική περίοδο. Διότι, όπως είδαμε, ζούμε σε ένα πραγματικό κόσμο. Δεν εφευρίσκουμε καταστάσεις. Έχουμε ήδη μια ετικέτα στα μαγαζιά. Ό,τι και να κάνουμε, θα υπάρξει μια μετάβαση προς ένα νέο μοντέλο. Πρέπει λοιπόν να το δούμε αυτό, τη μετάβαση. Μπορεί να ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν καινοτομίε, άρα τα πράγματα θα κινηθούν και σιγά σιγά θα υπάρξει μια εξέλιξη. Η μετάβαση αυτή έτσι κι αλλιώς λοιπόν θα γίνει. Αυτό που εμείς θελήσαμε να κάνουμε είναι να το λάβουμε αυτό υπόψη. Ακούστηκε ένα νούμερο, περίπου 72% καταλαβαίνουν το μοντέλο AG. Αυτά είναι τα προϊόντα που πουλιώνται σήμερα. Αυτή μετά από λίγο θα πρέπει να αλλάξει την τάξη, την ταξινόμηση και μια κατηγορία Α μπορεί να γίνει σε, ας πούμε, μετά από μερικά χρόνια. Τότε αυτοί ξαφνικά εγκαταλείπουν το πλοίο και έχουμε μόνο 19 ή 27% και 14% μόνο των ανθρώπων που υποστηρίζουν αυτό το σύστημα. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο αριθμών για τη διαβούλευση κονσουλτιών. Συνεδρίασε η Επιτροπή για, για τα σήματα ετικέτες. Καλέσαμε όλους τους ενδιαφερόμενους. Είχαμε ανταλλαγή ε, ταχυδρομικών στοιχείων κλπ. Ίσως ο κάθε ενδιαφερόμενος δεν πέτυχε αυτό που ήθελε. Οι βιομήχανοι δεν μίλησαν, αλλά και αυτοί ζήτησαν ορισμένα πράγματα, άλλου είδους ερωτήσεις θα μπορούσαμε να είχαμε θέσει ερωτήσεις πολύ πιο ενοχλητικές εντό εισαγωγικών στο ερωτηματολόγιο. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσει ζήτησαν και βάλαμε την τελευταία ερώτηση στο ερωτηματολόγιο. Δεν είναι δική μα πρόταση. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσει ζήτησαν και αποσύραμε την έννοια τη τιμή από το ερωτηματολόγιο. Γιατί επηρεάζει η τιμή τι επιλογέ. Λάβαμε υπόψη τι απόψει όλων όχι βέβαια 100% της απόψης του καθενός, διότι τότε δεν θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε μια τέτοια κατάσταση. Πάντως, τα περισσότερα τα λάβουμε υπόψη. Χρονολογία, ελήφθη υπόψη. Το μέγεθος των γραμμάτων, ελήφθη υπόψη. Προτείναμε μια επιπλέον ετικέτα, πέρα από την ενέργεια, να πούμε προσοχή, αυτό είναι μια παλιά ετικέτα ή προσοχή, αυτό είναι μια καινούργια ετικέτα η ετικέτα κατά τη γνώμη μας έπρεπε να αρκεί από μόνη της. Βέβαια μπορούμε ακόμα περισσότερο να ε, κάνουμε ακόμα πιο σαφείς τις πληροφορίες για τα ελαστικά αυτοκινήτων. Καλή ερώτηση. Γιατί προτείναμε μια ετικέτα ΑΖ για τα λάστιχα. Εμείς την ταξινόμηση την κάναμε έτσι ώστε η Α να είναι τόσο απαιτητική ώστε έχουμε κάμποσα χρόνια ακόμα μέχρι ότου οι κατασκευαστές να έχουν τα περισσότερα λάστιχα στην κατηγορία Α. Οπότε δεν προβλέπουμε να συμπλήψει αυτή η α ή α γιατί εξ αρχής η κλίμακα συνετέθη με αυτόν τον τρόπο. Δεν προδικάσαμε δηλαδή τις εξελίξεις αν μετά θα είναι α συν ή α Τα πράγματα παραμένουν ανοιχτά όσον αφορά τα ελαστικά αυτοκινήτων. Τώρα, κάτι άλλο. Θα πρέπει η ετικέτα να είναι κατανοητή. Φυσικά. Ακούσαμε το α-μείον, ο κόσμος δεν θα το καταλάβει. Ίσως το αζέν είναι πιο κατανοητό. Κάποιος που έχει ένα α που είναι λιγότερο καλό από το β, κακή επιλογή. Πρέπει να δει κανείς το σύνολο των προβλημάτων διότι αν αρκιστούμε στο άλλο ζ, δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. Θα ήταν πάρα πολύ απλό να κρατήσουμε το α, ζ. Το πρόβλημα είναι ότι τα πράγματα αλλάζουν και πάμε προς νέες γενιές. Αυτή η μετάβαση είναι δύσκολη. Και ελπίζουμε με τα στοιχεία αυτά εδώ θα βοηθήσουμε να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις. Και σας πληροφορώ ότι μέχρι αύριο θα είμαστε σε θέση να σας δώσουμε λεπτομέρειες όλα τα στοιχεία και όλα τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν σε όλους σας. Ο καθένας έτσι θα μπορεί να δει σε λεπτομέρειες του τι έγινε και να καταλήξει σε κάποιο πόρισμα. Ευχαριστώ κύριε Μάρα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα μόνο να σας υποβάλω δύο σύντομες σκέψεις αν θα μπορούσε να είναι εναλλακτική λύση το α συν συν ε, για να λυθεί το πρόβλημα. Ξέρουμε επίσης από τους καταναλωτές ότι δεν το καταλαβαίνουν πολύ καλά ε, αν υπάρχουν κατηγορίες πάνω από την α, α συν, α συν συν, αλλά θα πρέπει να συζητηθεί αυτό στην Κανονιστική Επιτροπή. Μπορούμε να το συζητήσουμε ως εναλλακτική λύση με την προϋπόθεση ότι θα ισχύσουν τα εξής. Πρώτον, πάνω από την α να μην υπάρχει άλλη κατηγορία αν δεν ε, δικαιολογείται τεχνολογικά γιατί έχουμε ε, ψυχία πλέον μόνο α, α συν και α2 συν και από το β μέχρι το g δεν έχεις καμιά συσκευή. Τι να την κάνω τότε την κλίμακα. Ε, θα πρέπει βεβαίως όταν κάποιοι είναι πρωτοπόροι να δαμηθούν και να πάρουν ένα συν, ένα πόντο επιπλέον αλλά εφόσον υπάρχει μόνο τεχνολογική δικαιολογία και ανάγκη. Και ένα δεύτερο για το α συν δεν θα πρέπει τα συν, στα ε, σταυροί να αυξηθούν ε, ε, στο δίνεκες. Απάνω από τρία συν δεν έχουν νόημα, δεν θα καταλάβει τίποτα ο καταναλωτής. Και όταν φτάσουμε στα τρία συν τότε χρειάζεται αναθεώρηση. Γιατί αν έχουμε πάνω από 7 κατηγορίες δείχνει ότι Υπάρχει πολύ μεγάλη διακύμανση ε, στην αγορά, μεγάλη γκάμα προϊόντων και μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο καλύτερο και στο χειρότερο προϊόν. Ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να διαλέγει ανάμεσα στα καλύτερα. Ε, ρωτήθηκε κάτι αν καταλαβαίνει ο καταναλωτής. Φαίνεται να λέει η Κομισιόν ότι δεν καταλαβαίνουν το α έως g οι καταναλωτές και δεν το προτιμούν υπήρχε μία διαφάνεια με ψυγεία κατηγορία C, παλιά και νέα, με διαφορετική αποδοτικότητα και 59% των καταναλωτών διάλεξαν το πιο οικονομικό προϊόν. Δεν έχουμε μελετήσει τα στοιχεία σε βάθος, δεν μπορούμε προς το παρόν να ε, πούμε περισσότερα. Χρειάζεται ανάλυση σε βάθος για να καταλάβουμε και εμείς από τα συμπεράσματα της έρευνας τι θα βγάλουμε. Ευχαριστώ. Η συνάδελφό σας κυρία Κλεμόλα πολύ σύντομα. Παρακαλώ σκεφτείτε και το χρόνο όμως. Ευχαριστώ. Επανέρχομαι σε ορισμένες ερωτήσεις και θέλω να προσθέσω μερικά πράγματα που αφορούν την εκπαίδευση των, ε, του, του, κλάδου πωλήσεων, του λιανικού κλάδου δηλαδή, από πλευράς καταναλωτών. Τι μπορούν οι, οι καταναλωτές να κάνουν. Ε, βεβαίως ε, πρέπει και εμείς να ενημερώνουμε τον καταναλωτή και ο καταναλωτής με τις επιλογές του κατευθύνει, δείχνει στο βιομήχανο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάντοτε ενήμεροι των εξελίξεων στην αγορά καθημερινά. Ποιες είναι οι, ανώτα, οι ανώτατες κατηγορίες σε ποιες μάρκες ε, στις συσκευές ε, η κλειστή κλίμακα A ε, to G την έχουν υποστηρίξει το λιανικό εμπόριο στη Γαλλία και στο Ενωμένο Βασίλειο διότι μα είπαν ότι του διευκολύνει ιδιαίτερα για να είναι ενήμεροι συνεχώ ποια είναι η ανώτατη κατηγορία και να μπορούν να την προσφέρουν. Όσον αφορά τώρα τι συζητήσει και τι διαβουλεύσει με τι ενώσει καταναλωτών, συμφωνώ με τη συνάδελφό μου από τη μη κυβερνητική οργάνωση, ασφαλώ στην φάση προετοιμασία του ερωτημολογίου συζητήσαμε με πολλές ενώσει καταναλωτών. Δυστυχώς πολλές επιφυλάξεις και ανησυχία μας δεν ε, λήφθησαν υπόψη. Περιμένουμε τις, τα τελικά στοιχεία και τα συμπεράσματα της έκθεσης της Κομισιόν για να ολοκληρώσουμε και τη δική μας μελέτη. Βεβαίως λάβαμε υπόψη το κόστος κατασκευής. Είναι σαφές ότι μια ε, σαφής ετικέτα μια εύκολη ε, ταυτότητα επιφέρει ένα κόστος. Το, το καινούριο σύστημα αξιολόγησης και ετικετοποίησης θα επιφέρει μεγαλύτερο κόστος από το καθημερινό κόστος ε, ενημέρωσης που κάνει το κατάστημα έτσι κι Ο κύριος Φαλτσόνη. Ευχαριστώ πρόεδρε ακούγοντας, ε, παρακολουθώντας αυτή τη συζήτηση, ε, διαμορφώνω την άποψη ότι υπάρχει μια διχογνωμία μεταξύ βιομηχανίας και καταναλωτών. Αλλά άμα κάνεις ένα κύκλο σπουδών ε, marketing, είναι ακριβώς η προτεραιότητα του καταναλωτή. Ο καταναλωτής είναι ο βασιλιάς, έτσι βασιλεύει στην αγορά. Πώς μπορούμε τώρα αυτό το μάθημα, αυτή την ε, αλήθεια να την ε, εφαρμόσουμε στην πραγματικότητα. Τα, ό,τι κάνουμε πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία, στην πραγματική κατάσταση. Ο καταναλωτής δεν θα καταλάβει το α μείον 20, 30, 40, οτιδήποτε θα καταλάβει το α έως g, το α έως ε, το α έως σίγμα ταφ, ε, την κλειστή κλίμακα, Ποια είναι τα στοιχεία, τα στοιχεία στα οποία βασιστήκατε ε, για να προτείνετε τις, ναι, τις αλλαγές. Ποιες είναι η απόφαση, η επιστημονική βάση δηλαδή της, της πρότασης. Ευχαριστώ κύριε Ποδηματά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε είναι αρκετά δύσκολο να εξαχθούν ορισμένα κοινά συμπεράσματα από αυτή τη συζήτηση Ακούσαμε τα επιχειρήματα όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών. Σε μεγάλο βαθμό αυτά τα επιχειρήματα τα γνωρίζαμε. Υπάρχει βεβαίως το καινούργιο στοιχείο που είναι η έρευνα της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακούσαμε τα βασικά συμπεράσματα από τον κύριο Αντρέ Μπριζάρ όπως όμως είπε και ο ίδιος, δεν έχουμε ακόμα δει τα πλήρη ερωτηματολόγια και τα πορίσματα της έρευνας για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια πλήρη εικόνα. Υπάρχει επίσης το στοιχείο ότι η μελέτη η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταλήγει σε διαφορετικά συμπεράσματα από αυτά στα οποία καταλήγουν μια σειρά από εθνικές μελέτες, έρευνες, πανεπιστημίων, καταναλωτικών οργανώσεων Ινστιτούτων και δεν νομίζω ότι ε, αρμόζει να επιχειρήσουμε εδώ να λύσουμε το θέμα της αξιοπιστίας της μιας μελέτης σε βάρος μιας άλλης. Εκείνο το στοιχείο ωστόσο που θα ήθελα να υπενθυμίσω είναι ότι εάν υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μια επιφυλακτικότητα που διατυπώθηκε από ορισμένου συναδέλφους ως προς την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από την ε, πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μια καχυποψία που εδράζεται στο γεγονός ότι τον περασμένο Απρίλιο επιχειρήθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί μια μελέτη επιπτώσεων ή μια έρευνα σαν αυτήν για την οποία κουβεντιάζουμε σήμερα, τα βασικά της συμπεράσματα, να αλλάξει η ενεργειακή σήμανση και να περάσουμε στην ε, ανοιχτή κλίμακα A-20-40 για τις τηλεοράσεις και τα ψυγεία. Και αυτό ήταν ε, ένα στοιχείο που συγκρατήθηκε από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με αυτή την έννοια και με αυτή την έννοια ε, υπήρξαν σκέψεις, ενστάσεις ως προς το αν μέσω αυτής της μελέτης υπήρξε πραγματικά η πρόθεση να επιλέξουμε την καλύτερη δυνατή σήμανση εκείνη που προκρίνουν οι καταναλωτές χωρίς ε, να έχουμε κάποια προτίμηση. Εκείνο που θέλω να διαβεβαιώσω είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την πλευρά του, το οποίο έχει δώσει μια σαφή κατεύθυνση σε πρώτη ανάγνωση, δεν έχει κανένα συμφέρον από την επιλογή της μίας ή της άλλης ενεργειακής σήμανσης. Και εκείνο που θέλω να τονίσω ε, είναι ότι από την ε, πλευρά όλων μας εκείνο που έχει σημασία είναι αυτό που είπα και στην αρχή ότι η ενεργειακή σήμανση ήταν ένα success story για την Ευρώπη για 17 χρόνια και ότι το βασικό κριτήριο, ο βασικός γνώμονας από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσει να είναι και το επόμενο διάστημα. Και μια μικρή ε, επισήμανση επ' αυτού ε, στόχος μας είναι η ενεργειακή σήμανση να αναγνωρίζεται από όλους τους ευρωπαίους πολίτες από όλους τους ευρωπαίους καταναλωτές από άκρου σ' άκρου της ευρώπης τόσο στο βορρά όσο και στο νότο στα νέα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης από τις πιο ευάλωτες κοινοτικές ομάδες από τα χαμηλότερα μορφωτικά στρώματα. Η ενεργειακή σήμανση δεν είναι ένα σοφιστικέ εργαλείο για να απευθύνεται μόνον στους πλέον ε, μορφωμένους ή στους πλέον συνειδητοποιημένους καταναλωτές. Η ενεργειακή σήμανση είναι ένα εργαλείο για να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο τη συνοχή στην ευρωπαϊκή επικράτεια και την ισόρροπη προώθηση Τη εξοικονόμηση ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και για την συμμετοχή σας και για τα σχόλιά σας σε αυτή τη συζήτηση και εκφράζω με τη σειρά μου, με τη βοήθεια των εξαιρετικών σκιωδών εισηγητών, ότι θα μπορέσουμε ε, να καταλήξουμε σε μια, στην καλύτερη δυνατή επιλογή, σε μια επιλογή που πραγματικά να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των καιρών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ μαζί σας και τους προσκεκλημένους αλλά εξ ονόματος όλων σας ιδιαίτερα την ισχύτρια την κυρία Ποδηματά πάρα πολλή δουλειά παραμένει λίγη δουλειά ακόμα ευχαριστώ πάρα πολύ ευχαριστώ πολύ εδώ ολοκληρώνεται αυτό το θέμα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα 2-3 λεπτά και θα συνεχίσουμε με το επόμενο θέμα ευχαριστώ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 θα διακόψουμε τις πάρα πολύ σημαντικές συνομιλίες που οπωσδήποτε πρέπει να κάνετε στην αίθουσα και τις αναβάλουμε είτε για άλλη χρονική στιγμή είτε εκτός της αιθούσης, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα προσκεκλημένο. Ich darf in Ihrer aller Namen Εξ ονόματος όλων σας καλωσορίζω θερμά τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κοινοτομίας και Τεχνολογίας, κύριο Μάρτιν Σιούρμανς. Σούρμανς το λέω στα γερμανικά, είναι λάθος. Πώς το προφέρετε, Σιούρμανς. Ο κύριος Βανίστε Ρόι μπορεί να τα πει καλύτερα από μένα. Για έλα να προεδρεύσεις λίγο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, θα προσπαθήσω όσο μπορώ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ που βρήκατε το χρόνο να έρθετε. Είμαστε πάρα πολύ περίεργοι να μάθουμε τι συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Έχουμε συζητήσει εντατικά εδώ και τσακωθήκαμε κιόλα για το εάν και πώς και πού και κατά πόσο πρέπει να ιδρυθεί το Ίδρυμα αυτό. Βλέπετε συναδέλφους εδώ που έχουν πολύ μεγάλη περιέργεια να μάθουν. Έχετε το λόγο. Καλώς ορίσατε κύριε Σιούρμαντς. Ευχαριστώ κύριε κυριε στα αγγλικά. Θα έλεγα καλημέρα στα αγγλικά. Μ' ακούτε καλά. Ωραία. Είναι μεγάλη χαρά που, για μένα που βρίσκουμε εδώ σήμερα για να σας ε, εξηγήσω πού σε ποιο σημείο βρισκόμαστε με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομία και Τεχνολογία, το EIT, γιατί πολλοί από εσά και καινούργια μέλη και ίσω καλό θα ήταν να κάνω μια γενική εισήγηση καταρχά στο τι είναι αυτό το ε, ίδρυμα, το αυτό το Ινστιτούτο. Είναι ένα καταλήτης για να ξεκινήσει και να προωθηθεί η αλλαγή, η στις, ε, ε, στις ευρωπαϊκές κοινότητες στον τομέα της καινοτομίας, ε, του δυναμικού και των, των επιπτώσεων. Θα επανέλθω στο δυναμικό στο θέμα του δυναμικού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα θεσμικά όργανα δηλαδή καταβάλουν προσπάθειες για να αυξηθεί το δυναμικό. Το EIT ε, εστιάζεται ε, στις επιπτώσεις της, και, της καινοτομίας βασικά. Ε, ξεκινήσαμε τη λειτουργία μας, μάλλον υιοθετήθηκε η ίδρυση του Ινστιτούτου σε 11 Μαρτίου του 2008 ως ανεξάρτητο κοινοτικό όργανο. Πιστεύω ότι είμαστε το πρώτο Ινστιτούτο αυτού του συγκεκριμένου τύπου. Δηλαδή, ανεξάρτητο στη λήψη αποφάσεων, από την άλλη πλευρά βεβαίως υπόλογο σαφώς στην Ευρωπαϊκή ε, ε, Κομισιόν. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι κάτι το εξαιρετικό το οποίο δεν το έχετε δει να γίνεται πολλές φορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, καλύπτουμε και τις τρεις πλευρές ε, του γνωστικού τριγώνου, ε, της καινοτομίας, ε, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, στο, επιχειρησιακή καινοτομία, θέλετε, επιχειρήσεις και καινοτομίες Είχαμε οργανώσει μία συνάντηση στο Γκότεμπορκ και μας, μας ρώτησαν ποιες από τις τρεις πτυχές είναι πιο σημαντικές για το Ινστιτούτο σας και εγώ απάντησα ότι και οι τρεις είναι ισότιμες στη σημασία διότι όλοι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι χρειάζεται πρωτοπορία, χρειάζεται καινοτομία. Η καινοτομία δεν ε, αρχίζει, δεν υπάρχει μόνο στην ε, εκπαίδευση και στην έρευνα ή στις επιχειρήσεις. Παντού, παντού η καινοτομία υφίσταται σαν στοιχείο. Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι με στο δίκτυο, στον ιστό της καινοτομίας καλύπτουμε και τις τρεις πλευρές Έχουμε λοιπόν ε, λάβει μια συγκεκριμένη εντολή ε, να, οργανώσουμε το Ινστιτούτο μας με μια ελαφρά, όχι πολύ ε, βαριά και περίπλοκη δομή σε δύο βαθμίδες. Είμαι καταλαβαίνω απόλυτα την ανάγκη της απλούστευσης ότι τα πράγματα πρέπει να τα οργανώνουμε με τρόπο απλό και έχουμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Καινοτομία και Τεχνολογία. έχουμε με 18 μέλη ένα θαυμάσιο διοικητικό συμβούλιο το οποίο υποστηρίζεται από το, την έδρα μας, την έδρα του Ινστιτούτου στη Βουδαπέστη. Επίσης, καλό είναι να σας ενημερώσω ότι ο Γεράρντε Ναζάλ όπως αποφασίσαμε πριν από δύο εβδομάδες, θα είναι ο διευθυντής του EIT. Έχουμε λοιπόν πλέον και τη θέση του διευθυντού και τον κατάλληλο άνθρωπο. Αυτό, αυτή είναι η πρώτη βαθμίδα λοιπόν. Εν συνεχεία έχουμε την επιχειρησιακή ε, βαθμίδα, την επιχειρησιακή εφαρμογή. Μιλάμε για δύο-τρεις ε, μόνο ε, κοινότητες καινοτομίες, καινοτομιακής γνώσης που θα καθοριστούν μέχρι το 2009. 309 εκατομμύρια είναι το budget μας. Είναι αρκετά μετριοπαθές θα έλεγα για να καλυφθούν αυτές οι κοινότητες. Τώρα θα σας παρουσιάσω τις κατευθυντήρες μας γραμμές στη δουλειά μας. Τι, τι θα κάνουμε, τι κάνουμε από απόψεως εργασίας. Καταρχάς, ε, εστιάζουμε ιδιαίτερα την προσοχή μας στην, ε, στο leadership, στην, ε, στο να είμαστε επικεφαλής. Όπως αποφασίσαμε πέρσι το Σεπτέμβριο, είπαμε ότι μέχρι το 2010 θα έχουμε αναλάβει, θα είμαστε επικεφαλής ε, πολλών ε, προγραμμάτων και εν συνεχεία θα μελετήσουμε τα διάφορα στοιχεία αυτών των προγραμμάτων τα οποία εμείς αναλάβουμε ως επικεφαλής. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα Η προκήρυξή μας ήταν, κάλυπτε μόνο 9 σελίδες. And I trust the intellect of the proposals. Ε, η προκήρυξη για την ίδρυση του οργανισμού και ε, αυτό επειδή ήταν πάρα πολύ σαφείς οι προτάσεις οι οποίες έγιναν και τις οποίες ε, θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Και συνεχεία θα, επανα... θα σας αναφέρω ένα μήνυμα που προέρχεται από τον πρόεδρο Ομπάμα, αλλά ε, το ιστορικό του είναι παλαιότερο. με μπερδεύει συνέχεια η Ευρώπη η οποία συνεχώς προβάλλει προσκόμματα και εμπόδια για το τι είναι δύσκολο να γίνει ότι υπάρχουν χίλιοι να κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε εκείνο και όπως είπε και ο Ομπάμα, yes we can. Δηλαδή, ναι μπορούμε. Εγώ αυτή την αντίληψη έχω, αυτή την γραμμή θα ακολουθήσω. Ναι μπορούμε. Και μπορούμε να παραδώσουμε και το έργο μας. Μπορούμε να κάνουμε και να παραδώσουμε αυτό που μας ζητάνε. Εν συνεχεία, ε, όπως σας είπα, εστιάζουμε, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην, ε, στις επιπτώσεις, στο αποτέλεσμα των καινοτομιών. Ε, μελετούμε το σύστημα εκπαίδευσης, ε, το, το, τον επιχειρηματικό τομέα, την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Δηλαδή εξετάζουμε όλες τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη αηφόρο ανάπτυξη, αλλαγή του κλίματος και το μέλλον των ε, τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη. Αυτά είναι τα στοιχεία κλειδιά. Ε, και εδώ άλλο ένας, σας είπα ότι και επαναλαμβάνω ξανά ότι δίνουμε σημασία στην επίπτωση των καινοτομιών στην ε, Κομισιόν ε, πολλά άλλα προγράμματα εξολύσσονται που έχουν σχέση με την καινοτομία, ε, τα, τα GITs, τα προγράμματα πλαίσιο και άλλα παρεμφερή, τα οποία βεβαίως είναι αλληλένδετα διότι ενισχύουν και αναπτύσσουν το δυναμικό που υπάρχει στην τεχνολογία και στην καινοτομία και ε, καταγράφουν και όλες τις εθνικές δραστηριότητε σε αυτόν τον τομέα. Πού είμαστε σήμερα, πού βρισκόμαστε. Το Διοικητικό Συμβούλιο άρχισε τη λειτουργία του 15 Νάτου 2008 και ολοκληρώσαμε την, ε, τον μειοδοτικό διαγωνισμό για τα KICS ε, ε, τις κοινότητες δηλαδή καινοτομία τον στις 27 Αυγούστου 2009 τα πρώτα, οι πρώτες δύο-τρεις καινοτομικές κοινότητες θα επιλεχθούν το Δεκέμβριο 2009 ε, βλέπετε τα πράγματα προχωράνε πολύ γρήγορα ο στόχος μας είναι τρεις τέτοιες κοινότητες τρία τέτοια kicks να εγκρίνουμε, να επιλέξουμε αν δεν μπορέσουμε να βρούμε τρία κατάλληλα θα επιλέξουμε δύο το θέμα είναι να είναι υψηλή ποιότητα. Εν συνεχεία θα προχωρήσουμε σε ένα εφταετές απλό πλαίσιο συμβατικό μέχρι το 2010. Εφτά ε, απλό ε, συμβατικό πλαίσιο και όλα, όλη αυτή τη διαδικασία ε, θα την κάνουμε πριν από τις προθεσμίες που, έχουμε, που έχουν τεθεί. Δεν νομίζω να χρειάζεται να σε εξηγήσω εδώ μέσα στο σώμα και σε αυτή την επιτροπή τη σημασία της καινοτομίας στην Ευρώπη και το πόσο υπολοιπόμεθα του, της παγκόσμιας κοινότητας. Είμαστε πίσω από την, ε, τον άλλο κόσμο. Όχι ότι δεν υπάρχουν αρκετές ενδιαφέρουσες ε, ε, περιπτώσεις στην Ευρώπη, ναι, βεβαίω. Πολλά ενδιαφέροντα πράγματα έχουν συμβεί και θα σα αναφέρω μερικά πρόσφατα γεγονότα του καλοκαιριού. Θα σα εξηγήσω καταρχά την μορφή, το format μέσα στο οποίο δουλεύουμε. Το οποίο λέγεται Commons. Είναι μια νέα ορολογία την οποία πιστεύω θα υιοθετήσετε κι εσείς. Ε, είναι το ηλεκτρονικό, η λεγόμενη ηλεκτρονική τεκμηρίωση, ηλεκτρονικό χαρτί. Εάν ήσασταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλατε να κάνετε ηλεκτρονικό χαρτί, electronic paper, δεν θα μπορέσετε να το επιτύχετε στις ε, Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί, διότι κάθε συστατικό του ηλεκτρονικού χαρτιού, είτε είναι η οθόνη, είτε κάποιο άλλο hardware, όχι μόνο κατασκευάζεται, αλλά σχεδιάζεται κιόλα στην Κίνα, στην Νότιο Κορέα και σε άλλα χώρες της Άπο Δηλαδή, αυτή η γεωγραφική περιοχή του κόσμου είναι αυτή η οποία τελικά έχει απλό, έχει όλο τον έλεγχο της, ε, του σχεδισμού και της ε, κατασκευής ο οποίος έλεγχος έχει φύγει από τα χέρια της Ευρώπης και εν μέρει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πολύ, ε, πολύ στο βιομηχανικό τομέα, στον κλάδο αυτόν, αργιούνται τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Όπως ξέρετε, πάρα πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες αναθέτουν τις εργασίες τους ή τμήμα εργασιών τους και της παραγωγής τους στην Κίνα, στην Ταϊλάνδη, στο Βιετνάμ. Τώρα λοιπόν με την οικονομική κρίση και με, την, ε, με το πρόβλημα του περιβάλλοντος ε, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πολύ και και η βιομηχανία αρχίζει και αλλάζει σιγά σιγά στάση και λέει ότι εάν μπορώ εγώ να έχω προμηθευτές από την Ευρώπη ας πάρω τους Ευρωπαίους προμηθευτές. Αλλάζει δηλαδή η προσέγγιση. Δεν είναι απαραίτητο ντε και να πάω στη Μανίλα για να βρω προμηθευτές. Βεβαίως ακόμα ε, υπάρχει η αμερικανική πλευρά η οποία κάνει την εξωτερική ανάθεση στο Μεξικό. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και τις δικές μας πηγές και να δούμε τι υπάρχει στο, στο δικό μας σπίτι. Μιλάμε για ενέργεια, μιλάμε για ε, δημογραφικά στοιχεία, μιλάμε για το περιβάλλον. Όλα αυτά σημαντικά στοιχεία για την κοινωνία μας. Άρα προσφέρονται και ευκαιρίες. Έχοντας περάσει πάρα πολλά χρόνια στην Κίνα, ε, πάρα πολύ καιρό τη ζωή μου στην Κίνα, θα έχω πολλά να σας πω για την εμπειρία μου αυτή και θα σας ε, αναφέρω μερικά παραδείγματα. Σήμερα κάθε μήνα ε, φτιάχνει ένα θερμοελεκτρικό εργοστάσιο το μήνα. Άνθρακα. Ε, με τεχνολογία από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ποια είναι η μόνη χώρα του κόσμου που έχει κάνει πείραμα με ε, πυρηνικό εργοστάσιο τετάρτης γενναίας, η Κίνα. Ποια είναι η μοναδική εταιρεία στον κόσμο που έχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ε, στέλνει και φτιάχνει και μπρίζες ηλεκτρονικές ε, για να φορτίζονται στη Σανκάη και στο Πεκίνο, η Κίνα. Εμείς μιλάμε, αυτοί δρούν. Αυτά όλα είναι αδυνηρά μηνύματα και καλό θα ήταν να επιταχύνουμε και να ε, έχουμε έτσι μαζική δράση και αντίδραση. Είναι υποχρεωτικό αυτό για την Ευρώπη. Και μία από τις πρωτοβουλίες αυτές είναι το δικό μας Ινστιτούτο. Αν θέλετε να συνεχίσετε επόμενη διαφάνεια. Ναι. Λοιπόν, ας πούμε λοιπόν δύο στοιχεία για περισσότερη καινοτομία στην Ευρώπη. Το δυναμικό είναι σημαντικό γιατί έχουμε αυτό το ωραίο πρόγραμμα της Λισαβόνας 2% και μετά συνεχίσουμε προς 3%. Είμαστε ακόμα κολλημένοι ούτε καν στο 2% λίγο πιο κάτω. Έχουμε χώρες που το βάλουν πολύ καλύτερα Ισραήλ, Σουηδία, Αυτά όμως γίνονται τώρα που μιλάμε και από εθνικές κυβερνήσεις και από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο εννοώ. Δηλαδή υπολογίζουμε στο ότι αυτό συμβαίνει. Αν δεν συμβεί, τότε δεν παίρνουμε στα σοβαρά την ευθύνη μας. Κυρίως κοιτάμε τι επίπτωση έχει η γνώση και να συνεχίσουμε μια νέα λίστα, νέες, νέα απασχόληση, νέοι άνθρωποι, αλλαγή κλίματος, μελλοντική κοινωνία, πληροφορίες, επικοινωνίας, βιώσιμη ανάπτυξη. Θα επανέλθω στις ε, κοινότητες γνώσης και επικοινωνίας. Εδώ μιλάμε όμως για κάτι που θα οδηγήσει σε μια νέα κοινωνία, νέα απασχόληση και ελπίζουμε κατά κάποιο τρόπο και ένα είδος έλεγχος στις αλλαγές του κλίματος. επόμενο διαφάνεια. Τι θέλουμε. Το είπα και πριν. Πρώτον, το να έχουμε το πλήρες δίκτυο καινοτομιών, που σημαίνει να υπάρχει μια, ένας συνδυασμός έρευνας ανάπτυξης καινοτομίας. Είναι πρόκληση για όλους μας. Δυστυχώς η καινοτομία δεν σταματάει στα σύνορα. Η καινοτομία επιβάλλει αλλαγές. Θα σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα από την Κίνα γιατί έχω επενδύσει πολύ κατά κάποιο τρόπο στη χώρα αυτή. Οι φοιτητέ σε μια σχολή βιοϊατρική του δίνουμε χρήματα στο τρίτο έτο για τη δική του δραστηριότητα και μερικοί φεύγουν και με master's degree αλλά έχοντα και μια μικρή επιχείρηση στα χέρια του, τελείω διαφορετικό στυλ. Κάτι τέτοιο θα έπρεπε να υπάρχει και στην Ευρώπη. Τρίτο, συντοποθέτηση ατόμων, collocation. Είναι μια πολύ προκένεια, δυσνόητη και εγώ ίδιος στην αρχή δεν την καταλάβαινα. Συντοποθέτηση εννοούμε ότι παίρνουμε ένα μεγάλο κομμάτι της αλυσίδας της καινοτομίας σε ένα τοπικό κέντρο. Μπορεί να είναι ένα υπερεθνικό κέντρο, μπορεί να υπάρχουν πολλοί εταίροι, αλλά είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένο έτσι ώστε οι άνθρωποι στο κέντρο αυτό μιλάνε μεταξύ τους η ροή της γνώσης είναι συνεχής μπορεί να είναι επιχειρηματία, ένας ειδικό στην τεχνολογία, ένας φοιτητής, ένας καθηγητής πανεπιστημίου είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό διότι λέμε να κάνουμε δίκτυα Οποιοδήποτε δίκτυο όμως στην Ευρώπη δεν θα έχει θετικό αποτέλεσμα ε, στην ε, βιομηχανία ή στην εκπαίδευση. Διότι αν δούμε στη Δύση τι γίνεται όσον αφορά την καινοτομία. Αναφέρομαι κυρίως στις Μένες Πολιτείες. Βοστόνη, έζησα στη Βοστόνη. Καταπληκτικά μέρη. Μετά έχουμε το Πεκίνο, Τσινγιάν, τη Σαγκάη. Μετά έχουμε άλλες περιοχές, Μπάγκαλορ, παραδείγματος χάρη, στην Ινδία. Δεν λέω να επιλέξουμε μία πόλη στην Ευρώπη και να το κάνουμε κέντρο. Λέω να επιλέξουμε τα καλά που έχουμε, γιατί έχουμε πολλά καλά σημεία, να τα φέρουμε όλα αυτά σε ένα συγκεκριμένο σημείο συντοποθέτηση, όπως το είπα πριν. Απλές και ελαφρές δομές και διαδικασίες μια στάση can do, γίνεται Επιτρέψουμε τώρα να αναφερθώ λίγο την έστρα στο επόμενο σημείο. Τι κάνουμε σήμερα στην Ευρώπη. Και σωστά. Ό,τι κάνουμε γίνεται σε ένα περιβάλλον πολύ ελεγχόμενο. Καλώς. Αν όμως θέλετε να περάσετε προς καινοτομία πρέπει να περάσετε από ένα ελεγχόμενο περιβάλλον σε ένα περιβάλλον που δίνει δυνατότητα σε κάποιον να κάνει κάτι. Η πρόκληση δηλαδή είναι να ισοφορήσουμε κατά κάποιο τρόπο από τη μια μεριά την ευθύνη που έχουμε και ταυτόχρονα να δώσουμε τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να βγουν από το καβούκι τους κατά κάποιο τρόπο και να ψάξουν αυτό που θέλουν. Ένα άλλο στοιχείο λοιπόν είναι να πάρουν μέρος οι βασικές βιομηχανίες, τα μεγάλα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη. Αυτό δεν ξεκινάει από το μηδέν. Έχουμε άριστα ταλέντα, άριστα Ινστιτούτα στην Ευρώπη. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Και παρεπιπτόντως αν δεν είναι ακόμα άριστα, δεν είναι πάρα πολύ καλά και πάλι μπορούν να ωφεληθούν από την κατάσταση αυτή. Επόμενη διαφάνεια. Γνώση, κοινότητες μάλλον γνώσης και καινοτομίας. ΚΙΚΣ, όπως το λέμε στα αγγλικά. Είναι ένας ευρωπαϊκός τρόπος δράσης αυτός. Πώς είναι δυνατόν να δημιουργηθούν αυτού του είδους οι κοινότητες γνώσης και καινοτομίας. Είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση στι αρχές του χρόνου με τον ΟΣΑ στο Παρίσι. Ο ΟΣΑ κάνει πολύ ωραίε εκθέσει για την καινοτομία και περί του πρακτέου κλπ. Αν δείτε τις παραμέτρους καινοτομία, οι εκθέσεις αυτές είναι πάρα πολύ καλές. Μιλάμε για 100 έως 200 συνιστώσεις. Η, η βιομηχανία δεν είναι καινοτομία έτσι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε το βασικό καύσιμο. Συγγνώμη, τις, τις λίγες βασικές παραμέτρους που χρειαζόμαστε και με βάση αυτές να κινηθούμε. Αν πραγματικά μιλάμε για την βιομηχανία, παραγωγή ή καλύτερα πανεπιστήμια, χρειαζόμαστε πρόσβαση σε αυτά τα τρία στοιχεία έρευνα, εκπαίδευση, βιομηχανία και στα τρία. Ε, θα σας μιλήσω για τις λίγες βασικές προκλήσεις, αλλά προηγουμένως θέλω να σας πω ότι αυτές οι κοινότητες κατά κάποιο τρόπο είναι ένα πείραμα. Αλλά είναι ένα πείραμα που κι εσείς ως ε, Επιτροπή και εμείς δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να αποτύχει. Γιατί αλλιώ θα σας έλεγα ποιος άλλος στην Ευρώπη μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Δεν γίνονται άλλες τέτοιου είδους προσπάθειες. Με τέτοιου είδους εστίαση. Πολλά στοιχεία και θα επανέλθω σε αυτά. Καταρχήν έλεγχος του τριγώνου της γνώσης στην πράξη. Σας όρισα τι είναι αυτή η κοινότητα. Είναι μια εταιρική σχέση με συνεργασία, ε, διορθωμένη νομικά και οικονομικά και μια συγκεκριμένη συμμετρία. Ποιοι είναι οι εταίροι του ΚΙΚ αυτού. Είναι η, τα στοιχεία του τριγώνου. Η συντοποθέτηση, την ανάφερα και πριν, είναι ένα μεγάλο κομμάτι του δικτύου καινοτομία από κοινού με την εγκύτητα, α το πούμε έτσι. Δηλαδή, αν θέλετε οι φοιτητέ να μιλάνε με του καθηγητέ, να μιλάνε με του επιχειρηματίε, να μιλάνε με άλλου, μην έρχεται, ε, έρθετε να μου μιλήσετε για ένα δίκτυο 500 χιλιόμετρων. Δεν έχει νόημα. σας θυμίζω ποια είναι τα προϊόντα τα οποία θέλουμε να έχουμε. Δημιουργία νέων επιχειρήσεων, να ε, ε, καλλιεργηθεί το επιχειρηματικό πνεύμα, δημιουργία απασχόλησης και οτιδήποτε άλλο έχει επίπτωση στην κοινωνία. Δημιουργία ε, νέων επιχειρήσεων, new business. Είναι κλειδί για μας αυτού του είδους η βιομηχανία. Και είναι διαφορετικό όταν μιλάμε για κλίμα, η ενέργεια ή το μέλλον της τεχνολογίας της επικοινωνίας. Επίσης κλειδί για μας είναι το μερικές φορές οι επιχειρήσεις δημιουργούν, προσπαθούν να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις. Από τις κλασικές βιομηχανίες προσπαθούν να δημιουργήσουν νέες. Και υπάρχει δυσκολία σε αυτό και γι' αυτό θέλουμε να τις βοηθήσουμε. Το δεύτερο Βλέπετε εκπαίδευση. Ξεκινάω από εκπαίδευση και ανάπτυξη για άτομα με επιχειρηματικό πνεύμα. Επιχειρηματιών δηλαδή. Στην Ευρώπη έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης και μπορεί να ανταγωνιστεί με οποιοδήποτε άλλο στον κόσμο. Ωστόσο, Κυρίως εκπαιδεύουμε για απασχόληση. Σπάνια εκπαιδεύουμε κάποιον να γίνει επιχειρηματίας, να γίνει εργοδότης. Μερικοί θα μας πούν γιατί δεν μπορείτε, δεν μπορείτε να εκπαιδεύσετε ένα επιχειρηματία, θα, μου έλεγαν. Νομίζω ότι αυτό δεν στέκεται, δεν νοηθεύει. ο, ο κάθε άνθρωπος έχει μια προκαθορισμένη δυνατότητα, αλλά μέσα στο πλαίσιο αυτό μπορεί να τονιστούν ορισμένες πτυχές και μπορούμε να βοηθήσουμε να υπάρξουν περισσότεροι επιχειρηματίες στην Ευρώπη και μέσα αυτά τα KICS θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Επόμενη διαφάνεια. Οι μερικές βασικές προκλήσεις. Πρώτο η αριστεία. Πολύ συχνά στην Ευρώπη μιλάμε για αριστεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα μου πείτε με ποιον συγκρινόμαστε και μετά σιωπή. Στην Ευρώπη έχουμε άριστες δραστηριότητες. Αυτό που δεν κάναμε είναι να τις συνθέσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ψηλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεύτερο, πρέπει να βοηθήσουμε τις συνεχείς εξελίξεις στην ανώτερη εκπαίδευση, να δράσουμε ως καταλήτης και στη διδακτέα ύλη και στις διδακτικές μεθόδους. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, όχι από την Κίνα. Το να μαθαίνει κανείς κάνοντας, πράττοντας, δεν είναι χαρακτηριστικό της Ευρώπης και μερικοί βιομήχανοι το έχουν ήδη αναγνωρίσει. Προσπαθούμε να του βοηθήσουμε. Συγγνώμη, μερικά πανεπιστήμια το έχουν καταλάβει, γιατί θα ήθελα να ασκηθεί αυτή η δραστηριότητα από τα πανεπιστήμια μα. Μετά υπάρχει η εκπαίδευση όσον αφορά το επιχειρηματικό πνεύμα. Και μετά φυσικά υπάρχει πλήρη εκμετάλλευση αυτού του πνεύματος μέσω εταιριών που υπάρχουν, μικρές, μεσές, νέες επιχειρήσεις, νέα μοντέλα, όλα να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις. Κάθε χρόνο, αν κοιτάξει κανείς, βλέπει μερικές καινούργιες επιχειρήσεις σε σχέση με την πληροφορική κλπ. Αλλά κοίταξα τη λίστα των 500 μεγαλύτερων και συμποθέσουμε ότι οι 100 καλύτερε αλλάζουν κάθε μερικά χρόνια. Κάθε τρία με τέσσερα χρόνια αλλάζει αυτή, η λίστα των 100 πρώτων. Πόσες από τις νέες επιχειρήσεις που ανεβαίνουν στις 100 είναι ευρωπαϊκές. Πολύ λίγες. Αυτό μας δείχνει ότι όσον αφορά μοντέλα νέων επιχειρήσεων Δεν είμαστε και πολύ δημιουργικοί. Υπάρχει έρευνα τεχνική, τεχνολογική και μη τεχνολογική που, που οδηγεί σε πλήρη εκμετάλλευση ευκαιριών καινοτομία. Και εδώ ένα παράδειγμα. Πολλοί με τους οποίους συζητάμε στην Ευρώπη μας λένε έχουμε ένα σωρό εφευρέσεις γιατί συζητάμε για καινοτομίε. Άλλο εφεύρεση, άλλο καινοτομίε. Η εφεύρεση είναι ένας από πολλού τρόπου να έχει καινοτομίε. Οι Κινέζοι έγιναν γνωστοί και θα είναι πρώτοι στον κόσμο με καινοτομίε, με απομιμήσει σε καινοτομία. Η Νόκια και άλλες εταιρείες το χρησιμοποιούν αυτό. Υπάρχει καινοτομία που κινείται μέσω της ε, προσφοράς. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δηλαδή, ναι, είμαστε υπέρ τη βασικής έρευνα, αλλά πρέπει να δούμε και την καινοτομία που στηρίζεται στην τρέχουσα τεχνολογία και πώ θα το επιταχύνουμε αυτό. Αυτό εννοώ. Σα είπα ότι έχουμε ένα πολύ καλό δυναμικό στην Ευρώπη. Δεν είμαι απεσιόδοξο. Έχουμε καλά ερευνητικά κέντρα, τεχνολογικά κέντρα, ισχυρή βιομηχανία, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι όλοι αυτοί να συγκεραστούν κατά κάποιο τρόπο σε υπερεθνικά κέντρα που θα δώσουν πανευρωπαϊκές ευκαιρίες. Επόμενο slide. Κέντρα συντοποθέτησης είναι το πιο ακαθόδες θέμα σε σχέση με τις προτάσεις για τα ΚΙΚΣ. Στις συζητήσεις που έχουμε προεισαγωγικά βλέπουμε ότι η πραγματική μάχη πρέπει να δοθεί εκεί. Πιστεύω απόλυτα. Και έχω πολλούς φίλους και από τη βιομηχανία που λένε το ίδιο. Η έννοια ότι η γνώση κινείται μέσω του χαρτιού είναι ξεπερασμένη. Δηλαδή, η γνώση πρέπει να ρέει μέσω των ανθρώπων. Καλό να υπάρχουν φοιτητέ και κάποιο να κάνει μια επιχείρηση. Έτσι, αυτό είναι το σωστό. Μετά έχουμε το IPA, μια άλλη ενδιαφέρουσα ιστορία. Βέβαια, εδώ στην κοινότητα μερικοί περιμένουν από εμά να λύσουμε αυτού του είδου τα προβλήματα τη Ευρώπη. Αυτό δεν έχει και νόημα γιατί εμείς απλώς είμαστε μια ομάδα που διευκολύνει. Εμείς συνεργαζόμαστε με τα ΚΙΠΣ να υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική για όλους τους ενδιαφερόμενους με κίνητρα. Ήδη πολλοί από αυτούς ήδη ασχολούνται με τα θέματα αυτά, γι' αυτό δεν υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνία, δεν ξέρω, ίσως να ήταν μια καλή ιδέα. Γιατί εμείς μπούμε σε αυτό, θα καθυστερήσουμε για πάρα πάρα πολλά χρόνια. συζητώντας με Κινέζους και Αμερικάνους μου είπανε ότι Πρέπει να υπάρχει περισσότερη ορατότητα. Πρέπει λοιπόν το IT να χρησιμοποιηθεί περισσότερο για μεγαλύτερη ορατότητά μας. Επόμενο slide. Μερικά ειδικά σημεία. Αν θέλουμε αποτελέσματα, χρειαζόμαστε ηγεσία τύπου CEO. Δηλαδή, τι εννοώ. Αν έχετε ένα ε, επιχειρηματικό πρόγραμμα πρέπει να το μπορείτε να το μεταφράσετε σε πράξεις το business plan είναι το κλειδί με συγκεκριμένες επενδύσεις με συνεχή εστίαση στην επιχείρηση και αν διαβάσετε πολύ προσεκτικά το slide ένα παρακολουθούμενο επιχειρηματικό πρόγραμμα με στοχευμένες επενδύσεις με στόχο να δημιουργηθεί μέσω του προγράμματος αυτού νέα επιχείρηση. Μέχρι στιγμής έχουμε πάρει 20 προτάσεις για ΚΙΚ. Τις επιλέγουν μια Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και σύντομα θα γίνει η τελική επιλογή. Και το επόμενο ερώτημα είναι από εδώ και μπρος. Τι κάνουμε. Να σας πω αυτό που είπα και στην αρχή. Κατά κάποιο τρόπο πρόκειται για ένα πείραμα που προσωπικά δεν πρέπει να δεν θεωρώ ότι πρέπει να επιτρέψουμε να αποτύχει, αλλά είναι ένα πείραμα. Όταν κάνουμε ένα πείραμα, εγώ είμαι φυσικός και ξέρω Θέλουμε και πρέπει να μάθουμε από αυτό το οποίο θα παραχθεί. Τον Ιανουάριο δηλαδή θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία διδαχής. Τι πράξαμε σωστό, τι πράξαμε λάθος και πώς μπορούμε να βελτιωθούμε. Δεύτερο, υπάρχει βεβαίως καινοτομία στην Ευρώπη. Λίμωνο. Δεν έχουμε όμως πλέον ισχυρή την οτροπία ε, του αποτελέσματος, ή, αν δούμε τους κλάδους βιομηχανίας που ήδη λειτουργούν. Όπως σας είπα, αυτός ο ιστός καινοτομία έχει πολύ περισσότερες συνιστώσεις. Ακόμα και αν ένα ε, ε, ερευνητικό κέντρο κάνει φανταστικές εφευρέσεις, θα πρέπει να βγάζει και καινοτομία τελικά. Δηλαδή, σίγουρα θα επικεντρωθούμε σε αυτό, θα εστιάσουμε σε αυτό ε, τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνίας, αναγνώριση ε, αριστείας, ε, μια ακαδημία που να προαγάγει το επιχειρηματικό πνεύμα. Ζητώ συγγνώμη για αυτή την ορολογία. Δεν θα έπρεπε να είχα μιλήσει γι' αυτό. Χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν, αλλά δεν μ' αρέσει. Να σας εξηγήσω τι εννοώ. Η, η Ακαδημία Επιχειρηματικού Πνεύματος δεν είναι σχολείο είναι ένα σύνολο ανθρώπων ε, από τους οποίους ο καθένας είναι εξαιρετικός, άριστος επιχειρηματίας εντός Ευρώπης και πέραν των συνόρων της και μπορεί να βοηθήσει σε αυτά τα κέντρα συντοποθέτησης τους νέους επιχειρηματίες πολύ περισσότερο από την τοπική υποστήριξη, να δρούμε πιο γρήγορα δηλαδή. Και μετά ε, μιλήσαμε για άλλες μορφές ε, εκπαίδευσης Κάποια στιγμή το Ινστιτούτο μας θα πρέπει να σκεφτεί το θέμα των διπλωμάτων και των ε, πτυχίων. Γιατί σας μιλώ για την εκπαίδευση ε, στην επιχειρηματικότητα στα πανεπιστήμια. Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να ανταμείβονται καθηγητές, ομάδες, ακόμα και φοιτητές που προάγουν αυτές τις ε, έννοιες. Είναι μια προσπάθεια το Ινστιτούτο Καινοτομίας. Ήθελα ίσως να το πω από την αρχή αλλά σας το ξαναθυμίσω δεν είναι κάτι που θα έχει ίσους όρους παιχνιδιού όλοι ίσοι. Αν αυτό θέλετε ξεχάστε το. Είναι ένα εγχείρημα που προσπαθεί να βρει τα καλύτερα κέντρα στην Ευρώπη, να τα συνδέσει με καλύτερο τρόπο, να προχωρήσουμε με άλλη ταχύτητα και πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό σημαίνει ότι κάποια μέρη θα είναι κέντρα αριστείας και κάποια λιγότερο άριστα, έτσι, δεν όχι καλά. Ε, σίγουρα λοιπόν χρειαζόμαστε να κάνουμε πολλά για να ε, προάγουμε το επιχειρηματικό πνεύμα και τη δημιουργία ε, επιχειρήσεων. Να πω κάτι άλλο. Συνειδητά δεν μίλησα ακόμα για τη χρηματοδότηση όλου αυτού του εγχειρήματο. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Ε, αυτό που αποφάσισε να κάνει το Ινστιτούτο Καινοτομία είναι ότι χρηματοδοτούμε μόνο κατά 25% αυτέ τι κοινότητε καινοτομία. Τα ΚΙΚΣ. Επαναλαμβάνω. Θέλουμε τετραπλασιασμό ε, στη δική τους ε, συμμετοχή. Πολύ ασύνθιστο είναι αυτό, γιατί το λέω. Αν κάποιο θέλει να συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα, ωραία, μπράβο και θα σας φέρει πολλά θετικά, αλλά πρέπει να δεσμευτείτε και να δείξετε μια προσήλωση. Και εγώ δεν πιστεύω σε προσήλωση που συγχρηματοδοτείται κατά 50%. Το 25% είναι ε, υπέρ αρκετό και ευχαριστώ που μας ε, δώσατε μόνο 308 ε, για να πείσω και τους υπόλοιπους. Τα υπόλοιπα από πού έρχονται. Αλλά είναι αυτονόητα. Όταν συμμετέχουν ενδιαφερόμενα μέρη εκτό από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, υπάρχουν εθνικά προγράμματα περιφερειακά, να δώσουν και ήδη τη συμμετοχή του και τελικά θα βρεθούν τα χρήματα. Δεν είναι και τεράστιο το πρόβλημα. Αλλά ήδη από τότε τα 300 εκατομμύρια έχουν γίνει ένα δίσκομα δύο. Και μιλάμε για ενοτομία και κοινότητες μεγέθους που κάθε χρόνο θα ε, ε, χρειάζονται 50 με 100 εκατομμύρια. Συνεχίζουμε. Αν θέλει κάποιο να ε, έχει κάτι παγκοσμίας κλάσεως χρειάζεται και συγκριτική αξιολόγηση και βαθμολόγηση. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο από όλα αυτά που κάνει η Ευρώπη. Πάτε στον ΩΣΑ, τρώτε ένα καταπληκτικό δείπνο στο Παρίσι, στο πύργο του Άιφελ και συζητάτε γενικώ και τα λοιπά και καταλήγετε σε ε, εκθέσεις για βαθμολόγηση και για συγκριτική αξιολόγηση. Και τελικά αν θέλετε να το εφαρμόσετε δεν αξίζει αυτή η έκθεση. Ε, θα χρησιμοποιήσουμε όλες αυτές τις βασικές πληροφορίες που έχουμε από τον ΩΣΑ και από αλλού, αλλά τελικά ε, θα έχουμε πολύ συγκεκριμένα βαθμολο... μορφές για να προχωρήσουμε σωστά. Ήδη το κάνουμε αυτό εν μέρη, αλλά περιμένουμε και οι κοινότητες αυτές να συγκροτηθούν και να συνεννοηθούμε μαζί τους. Και τέλος, σίγουρα θα έχουμε μια στρατηγική ατζέντα καινοτομία για το Ινστιτούτο μας, για το μέλλον και πάλι από ό,τι καταλαβαίνετε αυτό θα χρειαστεί τη συμμετοχή όλων των εταίρων και παραγόνων εντός και εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό, είναι προφανές. Έρχομαι λοιπόν ε, στην τελευταία νομίζω, οι τελευταίες δύο διαφάνειες. βοηθήσουμε την υπάρχουσα βιομηχανία να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, ε, επιχειρήσεις, να βελτιώσουμε την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές και μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση κτλ. Υπό των όρων τώρα έρχονται οι όροι ότι θα αναγνωρίσουμε και θα δεχτούμε τις προκλήσεις αυτές στην Ευρώπη. Είμαστε πολύ καλοί στη συζήτηση και στην ανάλυση, αλλά δεν ε, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε αυτές τις προκλήσεις, δεν τις αποδεχόμαστε για να τις αντιμετωπίσουμε. Αν δεν υπάρχει επιχειρηματικό πνεύμα στην Ευρώπη, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε επιχειρήσεις να, να μαθαίνουμε από τις επιτυχίες μας και από τις αποτυχίες μας, να δώσουμε χρόνο στις κοινότητες αυτές να γίνουν παγκοσμίου ε, επίπεδου, χρηματοδότηση μέχρι 12 χρόνια, μακροπρόθεσμη και τέλος και νέες κοινότητες να συγκροτήσουμε καινοτομίε και χρειάζεται δράση και απόδοση και επιδόσεις. Είπαμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Can do. Ε, αν μπορούμε, ας τα κάνουμε τότε. Ε, χρειάζεται δράση πάντα. Αλλά η δράση να έχει και αποτέλεσμα. Αυτό για την Ευρώπη είναι ιδιαίτερο. Πολλές χώρες γύρω μας έχουν ε, πλέον αυτό το ύφος, αυτό το στυλ. Η Κίνα, η Ινδία. Πήγα στην Κίνα και τους μίλησα για το ε, κέντρο μας και ένας κύριος είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα αντίδραση πότε ξεκινάμε, τι σε ενδιαφέρει, πόσα λεφτά πρέπει να φέρω και πότε θες αποτελέσματα. Και παρακαλώ με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την οτροπία να λειτουργούμε και στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ähm, Ευχαριστώ. Σαφέστατα τα είπατε όλα αυτά. Ο κύριος Καβάλιο έχει το λόγο. Η κυρία Καβάλιο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και Πρόεδρε του EIT. Ε, το EIT είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία πράγματι ε, και μετά από μια δύσκολη αρχή ε, χαίρομαι που λειτουργεί ομαλά και απο, αποδοτικά. Καταρχάς θέλω να ρωτήσω πώς σε τι διαφέρει το EIT από το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο, το ERC και κατάλαβα βεβαίως ότι η πολιτική σας και οι στόχοι σας πρέπει να συμβαδίζουν ε, με τους στόχους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ε, πώς λοιπόν πιστεύετε ότι το EIT θα ταιριάξει μέσα στο νέο πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας ε, στο χρημα... υπολογισμό, στον προϋπολογισμό τον οποίο προτείνει η Κομισιόν για τις ε, καινοτομίες. Πώς ε, πιστεύετε ότι θα προσαρμόσετε τη λειτουργία του οργανισμού σας σε αυτό το πλαίσιο και πώς, πώς κρίνετε την καινοτομική στρατηγική στην Ευρώπη ο πρόεδρος της ε, Τελεστικής Επιτροπής ανέπτυξε τους στόχους ε, της επόμενης ε, θητείας του και επίσης είπε ότι έχει φιλόδεξους στόχους για όλους τους τομείς και της βιομηχανίας και της, του γεωργικού τομέα. Πιστεύετε ότι το δικό σας Ινστιτούτο μπορεί να συμβάλλει στις καινοτομίες αυτών των τομέων. Εν συνεχεία είπατε μάλλον στην αρχή ότι θα λειτουργήσετε ως καταλήτης ε, ως, φάρος των καινοτομιών ε, μειώνοντας ε, το κόστος και χρησιμοποιώντας ένα πολύ αποτελεσματικό μοντέλο. Θα συνεργαστείτε με άλλα δίκτυα, με πανεπιστήμια, με διάφορα άλλους οργανισμούς καινοτομία ε, για να αναβαθμίσετε το Ινστιτούτο σας. Ε, ε, με ποιου τρόπου πιστεύετε ότι θα προωθήσετε την καταλητική επίδραση του δικού σας Ινστιτούτου. Ο κ. Χατζημαρκάκης. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν έχω ερώτηση. Ένα σχόλιο θα ήθελα να εκφράσω. Το EIT είναι το δικό μας δημιούργημα, το δικό μας παιδί, διότι ε, πολύ γρήγορα ε, δημιουργήσαμε αυτό το Ινστιτούτο. Νομίζω ο πρόεδρος Μπαρόζο το 2005 ε, έθεσε τους πόρους και εν συνεχεία το 2008 λειτουργήσε. Είναι λοιπόν αυτό το δημιούργημά μας πραγματικά μια επιτυχία και είμαι ενθουσιασμένος που είδα την πραγματοποίησή του πρέπει να σας πω τι, τι μας ε, εντυπωσιάζει ιδιαίτερα και το λέω αυτό με μεγάλη περηφάνεια. Είναι αυτή η στρατηγική βάση ε, από την οποία ξεκινάει αυτό το Ινστιτούτο. Είμαστε βεβαίως ε, πρωτοπόροι στην ε, έρευνα και στην καινοτομία, αλλά μας έλειπε κάπως ο ευρωπαϊκός πατριωτισμός. Εντάξει, τα κράτη-μέλη είχαν τις δικές τους πολυσχηδείς και πολύπλευρες ερευνητικές προσπάθειες και καινοτομικές επιτυχίες. Αλλά το ευρωπαϊκό στοιχείο έλειπε, έλειπε το ευρωπαϊκό επίπεδο ε, και αναγνωρίσαμε ότι εμείς πρέπει στρατηγικά να μην χάσουμε από τα μάτια μας την καινοτομική αλυσίδα και πρέπει να την προωθήσουμε και να την προβάλλουμε. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που δεν ε, ορίζεται την καινοτομία και το, τις επιπτώσεις της καινοτομίας ε, με πολύ γενικούς όρους, αλλά λέτε τι θα ωφελήσει τον επιχειρηματικό κόσμο. Πού θα ανοίξουν καινούριες ευκαιρίες επιχειρηματικές. Από πού θα μπορέσουμε να κερδίσουμε περισσότερα, να βρούμε ένα οικονομικό όφελος. Δηλαδή αυτός ο επιχειρηματικός προσανατολισμός σας είναι σωστότατος και σας συγχαίρω για την ταχύτητα των ενεργειών σας πραγματικά λειτουργείται ε, ε, ταχύτατα. Εγώ δεν συμφωνώ ότι υπήρχαν δυσκολίε στην αρχή με την προλαλήσαντα συνάδελφο που το είπε. Εγώ πιστεύω ότι από την αρχή τα πράγματα ξεκίνησαν και εξελίχθηκαν πάρα πολύ καλά και γρήγορα. Το τρίτο κικ Πιστεύω η τρίτη καινοτομική κοινότητα θα πρέπει να ασχοληθεί, όπως είπατε, με το θέμα υγείας και διατροφής. Είναι μία, ένας ιδιαίτερος τομέας για μας τους Ευρωπαίους, διότι έχουμε διαφορετικές ε, προδιαγραφές και κάπως διαφορετικές προσεγγίσεις στον τομέα αυτών. Δηλαδή η πολύ στενή διασύνδεση του τρόπου διατροφής με τις επιπτώσεις επί της υγείας είναι θεμελιώδους σημασίας. Υπάρχει ακριβώς και μία μελέτη του STORE που θα σας τη στείλω. Στοα. Του που θα σας τη στείλω ε, και αναφέρεται σε αυτό το θέμα και επίσης άλλη μια κοινότητα καινοτομική θα επικεντρωθεί στην ε, κοινωνία της πληροφορικής. Ε, μην ξεχνάτε ότι εκτός από το επιστημονικό-τεχνικό προσωπικό πρέπει να υπάρχει και ένας ε, πνευματικός πλούτος, μια πνευματική ένα στοιχείο πνευματικής ιδιοκτησίας, βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ε, έχουμε θέματα προστασίας δεδομένων. Ε, μην ξεχνάτε λοιπόν η τεχνική πλευρά που καλύπτεται, αλλά μην ξεχνάτε και το πνεύμα. Τις θεωρητικές επιστήμες. Ο κύριος Λάμπαρτς. Ευχαριστώ κύριε Σιούρμαν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τοποθέτησή σας πραγματικά μεγάλο πάθος και το γυρίζω στα αγγλικά τώρα. Συμμερίζομαι και εγώ το πάθος και τον ενθουσιασμό σας. Συμφωνώ απολύτως και προσυπογράφω τα όσα είπατε για το κέντρο καινοτομίας ε, και για το τοπίο στο οποίο εγγράφεστε. Πρώτον, Έχετε βάλει τη σωστή εστίαση. Ως πράσινος βέβαια καταλαβαίνετε ότι θα το πω αυτό, ε, το κλίμα και η ενέργεια να είναι ε, στο κέντρο της στρατηγικής όπως και η τεχνολογία της πληροφορίας από την οποία προέρχομαι είναι μεγάλη ανάγκη. Ε, αλλά και χαίρομαι τον τρόπο που μας το ερμηνεύεται όχι μόνο ως ανάγκη αλλά και ως ευκαιρία και θα πρέπει να βλέπουμε και τους, ίδιους τους δύο όρους της εξίσωσης. Συμφωνώ όμως και με το επίγον του πράγματος που λέτε και μου αρέσει πολύ ο τρόπος που θέσατε την Ευρώπη απέναντι στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το έχω ξαναπεί εδώ στην Επιτροπή μας. Ε, κοιτάξτε τι έγινε στη διοίκηση Μπούς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν τετραπλάσιο το κεφάλαιο ε, κινδύνου για τις ανανεώσιμες από ό,τι στην Ευρώπη. Η Silicon Valley πριν από 20 χρόνια ε, ανθούσε από την πληροφορική, τώρα ανθεί από την πράσινη τεχνολογία σε μια χώρα που δεν πίστευε στην κλιματική αλλαγή τότε. Και είναι σωστό ότι θα πρέπει ε, να ξέρουμε τις ισχύει μας στην Ευρώπη και να ε, έχουμε και επίγνωση. Πολύ συχνά ε, βλέπω να ακούμε μια συγκατάβαση ότι είμαστε πρωτοπόροι στην πράσινη τεχνολογία και τι ωραίοι που είμαστε. Μην το δέσετε κιόλα αυτό. Είμαστε μπροστά σε πολλούς τομείς, αλλά πολύ γρήγορα που να χάσουμε αν δεν αντιδράσουμε γρήγορα. Γι' αυτό λέω ότι είναι επίγον το θέμα και σας υποστηρίζω απολύτως. Το τρίτο που με χαροποίησε ήταν αυτή η έννοια της συντοποθέτησης, co-location όπως το είπατε. Πριν από 20 χρόνια η εταιρεία μου ξεκίνησε την τηλεεργασία και τώρα βλέπουμε τι σημαίνει αυτός ο κατακαιρματισμός και που έχουμε σκορπίσει όλο τον κόσμο παντού στο σπίτι του. Ε, δεν υπάρχει αυτή η διάδραση και πραγματικά δεν ε, ρέει η γνώση όπως είπατε μεταξύ των προσωπών γιατί δεν συναντούνται. Σας ερωτώ τώρα για την καινοτομία. Καινοτομία ίσον τεχνολογία ε, ε, ε, το υπενηχθήκατε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και μια διαδικασία ολοκληρή και ο τρόπος με τον οποίο ενεργούμε και οργανώνουμε ένα επιχειρηματικό μοντέλο, business model για να το πω έτσι. Στο Ινστιτούτο σας αυτό το έχετε λάβει υπόψη και σε ποιο βαθμό. Πρέπει να το καταλάβω γιατί η τεχνολογία από μόνη της δεν θα λύσει το πρόβλημα. Το θέμα είναι πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε και πώς θα την αξιοποιήσουμε για να αλλάξουμε τα πράγματα. κατά την άποψή σας, ε, ποια είναι τα βασικά σημεία κλειδιά, τι τραβάει την προσοχή μας. Καταλαβαίνω το ενθουσιασμό για ένα έργο από την κοινότητα κτλ. Αλλά ε, σε όλη τη συζήτηση που γίνεται για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, βλέπω ότι πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν ένα πνεύμα ε, επαρχιώτικο εδώ χρειάζεται κοινοτική προσέγγιση, όχι ο καθένας ε, τα δικά του. Ε, αυτή την αντίληψη τη βλέπετε. Τα κράτη-μέλη δρούν ε, ξεχωριστά και δεν συμμετέχουν στις κοινοτικές πρωτοβουλίες. Μετά, τα χρήματα. Πού θα τα βρούμε. Καταλαβαίνω αυτό που είπατε για τη μόχλευση, γιατί όχι ότι ρέουν τα χρήματα και δεν μας νοιάζει. Θα πρέπει να βάλουμε το χέρι στην τσέπη και να δεσμευτούμε και να έχουμε και την ευθύνη. Αλλά ακούν αυτά τα χρήματα που έχουμε. αυτό με προβληματίζει. Και ένα τελευταίο θέμα, τα πνευματικά δικαιώματα. Όταν εγώ κάνω μια καινοτομία, είναι και κίνητρο αυτό να έχω ένα κέρδος. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ε, καμιά φορά χρησιμοποιούνται ε, ε, ως τροχοπέδι, γιατί όταν έχεις διπλώματα τεχνία, κάθεσαι και τα γλωσσάς και παίρνεις τα λεφτά σου και δεν προωθείς την καινοτομία και την εφαρμογή τους. Λοιπόν, είναι ευκαιρία για την Ευρώπη να ξαναγίνει τώρα βιομηχανική δύναμη και το, λέω συνειδητά αυτό, πρόκειται για τη βιομηχανία. Την έχουμε επεμπολίσει τη βιομηχανία και λέμε στην Ευρώπη τώρα είμαστε οικονομία υπηρεσιών. Εγώ πιστεύω ότι η ενέργεια, μεταφορές, η κλιματική αλλαγή είναι βαριά δραστηριότητα βιομηχανική και εμεί οι πράσινοι το καλωσορίζουμε γιατί έτσι έχουμε μια ισορροπημένη οικονομία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Γκίρεκ. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι, ότι το EIT από μόνο του είναι ένα παράδειγμα καινοτομίας. Άρα θετικό. Η καινοτομία χρειάζεται μια λειτουργούσα αγορά. Χρειάζεται πολύ καλή ποιότητα έρευνα, πολύ καλή ποιότητα. εκπαίδευση και ευελιξία όσον αφορά τον νόμο για τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Αυτοί οι τέσσερι παράγοντε βελτιώνουν την κοινοτομία. Το να φέρουμε την κοινοτομία στην αγορά το να φέρουμε την δημιουργικότητα στην αγορά είναι το θεμέλιο της οικονομίας μας. Για να γίνει αυτό πρέπει να κάνουμε μερικές αλλαγές. Πρώτον, λειτουργούσα αγορά. Λειτουργεί η αγορά. Είμαι όπως θα έπρεπε να έχουμε μια πιο καινοτόμα αγορά υψηλής ποιότητας έρευνα. Την έχουμε. Την εγγυάται το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Βέβαια δεν είναι στο ίδιο υψηλό επίπεδο σε όλες τις χώρες μέλη. Τρίτον, εκπαίδευση υψηλής ποιότητας. Πολλά πρέπει ακόμα να γίνουν στο μέτωπο αυτό. Αναφερθήκατε στην Κίνα, κύριο Μιλιτά. Η επιτυχία της εν μέρει έγινε στο ότι η εκπαίδευση Ιδιαίτερα η, η εκπαίδευση σε θέματα τεχνολογίας και θετικών επιστημών είναι υψηλότερο του επίπεδου. Στην Ένωση έχουμε ένα πρόβλημα προσπαθώντας να βελτιώσουμε αυτού του είδους την εκπαίδευση. Δεν έχουμε αρκετά άτομα που να ενδιαφέρονται. Τέλος, δημιουργικότητα και νόμος για τις ευρεσιτεχνίες. Πρέπει πρώτα να απαντήσουμε στο ερώτημα πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την καινοτομία. Θα ήθελα να σας κάνω και μια ερώτηση. Συζητήσαμε τη σύσταση του Ινστιτούτου σας. Στη συζήτηση αυτή ο κύριος Μπαρόσο ανάφερε αλλαγή του κλίματος, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και σύγχρονη τεχνολογία υπολογιστών ως τρία βασικά μεγάλα θέματα. Ο συνάδελφος πριν από μένα αναφέρθηκε στην αλλαγή του κλίματος. Ερωτώ λοιπόν, Θέλετε να δημιουργηθεί ένα μοντέλο αλλαγής του κλίματος με όλους τους παράγοντες μέσα που επηρεάζουν το κλίμα και όχι μόνο το διοξείδιο του άνθρακα ή θα δείτε σε τι βαθμό αυτές οι αλλαγές έχουν ήδη γίνει. Οι μελέτες σας, η έρευνά σας για την αλλαγή του κλίματος, τι κατεύθυνση έχουν. Πρόεδρος. Η κυρία Ριέρα Μαντουρέλ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω καταρχάς τον κύριο Σιούρμανς για την παρουσία του και να το συγχαρώ για το έργο του. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί του για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στην Ευρώπη και μετά όσα μας είπε για το μοντέλο του Ινστιτούτου που επιθυμούμε στην Ευρώπη να έχουμε που κατά τα άλλα το συζητήσαμε ευρύτατα στο Κοινοβούλιο και η αριστεία θα πρέπει να είναι στόχος πάντα στις εργασίες μας και όπως το είπε συμφωνώ με τα περισσότερα από όσα μας παρουσίασε. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του Ινστιτούτου και την αρχική πορεία. Μας είπατε από το 2008 τον Ιούλιο έχετε αποφασίσει για το Διοικητικό Συμβούλιο και επίσημα ξεκίνησε το Σεπτέμβριο τη λειτουργία του μετά ε, από τα εγγένεια της έδρας στη Βουδαπέστη. Εύκολα φανταζόμαστε τα ζητήματα που σας απασχόλησαν τους πρώτους μήνες εσάς και την ομάδα που σας πλησιώνει και τα στελέχη. Ε, για να αρχίσει τη λειτουργία του, να μπει το νερό στα βλάκια και να γίνουν ε, οι πρώτες προκηρύξεις για τις κοινότητες ε, καινοτομία ΚΙΚ. Και τώρα είναι το στάδιο της επιλογής αρκετά περίπλοκο και δύσκολο. Επιτρέψτε μου να σας κάνω συγκεκριμένες ερωτήσεις εγώ για το Ινστιτούτο. Η πρώτη έχει να κάνει ακριβώς με τη χρηματοδότηση. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, <clears throat> ήταν από τα θέματα που συζητήθηκαν περισσότερο στο Κοινοβούλιο. Γιατί δεν θεωρούσαμε υπεύθυνο να δημιουργήσουμε καινούργια δομή χωρίς την απαραίτητη και κατάλληλη χρηματοδότηση. Στις διαπραγματεύσεις ακούστηκαν διάφορα επιχειρήματα και μεταξύ αυτών ήταν η ίδια δυνατότητα που θα έχει το Ινστιτούτο για να κινητοποιεί πόρους, κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα, για την υποστήριξη της έρευνας μακροπρόθεσμα σε κάποιους τομείς και για να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου. Το είπατε κι εσείς και βεβαίως γνωρίζετε άριστα τον τομέα σας. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω, σας παρακαλώ, τι δράσεις θα αναλάβετε για να πείσετε, όπως είπατε, για να κινητοποιήσετε τη βιομηχανία πέρα από τους όρους και τις προϋποθέσεις ε, συμμετοχής στις κοινότητες καινοτομίας της ΚΙΚ. Και δεν είναι μόνο αυτό το στοιχείο της χρηματοδότησης. Πώς θα τους πείσετε να συμμετέχουν ως ε, φορείς, ως ε, εταίροι, ως πρωταγωνιστές στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Και επίση πάντα στη χρηματοδότηση θα ήθελα να μου πείτε παρακαλώ τι πιστεύετε για την πρόταση χρηματοδότησης. Περιγράψατε κάπως τη χρηματοδότηση αλλά δεν μας δώσετε την προσωπική σας γνώμη. Πρέπει να αλλάξει κάτι και αν ναι, εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεύτερη ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω. Ε, ενημέρωση και πληροφόρηση και επικοινωνία. Το είπατε κι εσείς. Είναι καινούριο φυσικά το Ινστιτούτο και θα πρέπει να γίνει γνωστό. Κάνατε μεγάλη προσπάθεια στην ενημέρωση, επικοινωνία, στο διαδίκτυο, έχετε ωραία ιστοσελίδα, με ενημερωτικά φυλάδια, ε, ευανάγνωστα στις 27 γλώσσες, ε, με σεμινάρια, ενημερωτικές ε, εκδηλώσεις για τους στόχους σας, τις προτεραιότητες σας, για την οργάνωση των κοινοτήτων, ΚΙΚΣ και στις διάφορες χώρες. Πολύ ωραία όλα αυτά. Αλλά το ένα είναι να ενημερώνει τον κλάδο, τα πανεπιστήμια, τους αποδέκτες σου, τις εταιρείε και άλλο διαφορετικό είναι η προβολή στην κοινωνία του Ινστιτούτου. Η γνωριμία από τον κόσμο. Εκεί χρειάζεται προσπάθεια. Θα πρέπει το Ινστιτούτο Καινοτομία να χρησιμοποιηθεί για να υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική συμμετοχή του, κόσμου, της κοινωνίας σε αυτά τα θέματα. Το MIT είναι γνωστό ε, στην Αμερική βεβαίως έχει μεγάλη πορεία, είναι πάρα πολύ γνωστό. Αλλά θα πρέπει και το δικό μας Ινστιτούτο να γίνει γνωστό στον κόσμο ευρέως. Και θα επιθυμούσαμε κάτι τέτοιο. Δύο πολύ σύντομε ερωτήσει. πρώτο γνωρίζουμε ότι έχει προκηρυχθεί διαγωνισμό για εμπειρογνώμονε σε διάφορους τομείς για να συμμετέχουν ως αξιολογητές αλλά και να υποστηρίζουν τις ε, κοινότητες ε, ε, καινοτομίας. Τι έχετε στο μυαλό σας, ποιο θα είναι το έργο με το οποίο θα τους επιφορτήσετε για την υποστήριξη στις κοινότητες αυτές. Και μια τελευταία ερώτηση. Όταν επελέγει η Βουδαπέστη ως έδρα του Ινστιτούτου, υπήρχαν και άλλες υποψηφιότητες διάβασα ότι οι πόλεις που δεν επελέγησαν έχουν τώρα το καθεστώς του κέντρου προώθησης του, του Ινστιτούτου. Τι σημαίνει αυτό, μπορείτε να μου εξηγήσετε, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Τόγια. Ευχαριστώ και εγώ για την παρουσίαση αυτή. Όπως και άλλοι συνάδελφοι και εγώ σας συγχαίρω για αυτά που είπατε και σε ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Με την έννοια ότι το Κοινοβούλιο, στο Κοινοβούλιο πρέπει να είμαστε κατά της δημιουργίας νέων δομών, νέων που πολλαπλασιάζονται ανεξέλεκτα κάθε μέρα. Πάντως το Κοινοβούλιο με πλειοψηφία ήταν υπέρ του να γίνει το Ινστιτούτο σας. Και έχει προσδοκίες σε σχέση με την ε, δραστηριότητα του Ινστιτούτου σας στο Κοινοβούλιο. Κάτι άλλο, η σημασία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και της πληροφορίας. Αναφέρεται συχνά ως διάσταση, αλλά η κατάρτιση δεν είναι απλώς εκπαίδευση, είναι η ανάπτυξη μιας τάσεις, δεν είναι μόνο επιστημονικές γνώσεις. Πώς στην Ευρώπη μπορούμε να δημιουργήσουμε μια στάση η οποία να είναι πιο καινοτόμα. Δεύτερο, για να καταλάβω κάτω, αυτή η συντοποθέτηση, collocation, τι ακριβώς σημαίνει. Φαίνεται να είναι μια νέα απάντηση, γιατί συχνά λέμε μπε στο δίκτυο, συνδέσουμε το δίκτυο, βάλε στο δίκτυο τα πράγματα, αλλά μιλώντας γενικά για δίκτυα, αυτό από μόνο του δεν δίνει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα στενή συνεργασία εννοώ. Εξηγήστε μας λίγο παραπάνω αυτή την έννοια, συντοποθέτηση, πως χρειάζεται μια συγκέντρωση των εμπειριών, του διαλόγου, μια συζήτηση ενώπιο σε Γιατί είπατε ότι με κόπο ε, να προωθήσετε αυτή την έννοια. Από τα κράτη-μέλη, η επιστημονική κοινότητα, τα κέντρα αριστεία σας απάντησαν θετικά και για τη σύσταση των ΚΙΚΣ, αλλά τουλάχιστον να, ξέρουν ότι υπάρχουν αυτά, ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα συντοποθέτηση. Δεν ξέρω αν η, στην Ιταλία είναι γνωστή αυτή η νέα πραγματικότητα. Ποια ήταν η απάντηση που σας δώσανε. Τέλος, επειδή είμαστε στην, ήδη στη φάση εφαρμογής, επειδή συμφωνούμε με τη θέση της Κομισιόν για το joint programming, δηλαδή την ανάγκη συντονισμού των προσπαθειών να πετύχουμε την κρίσιμη μάζα. Είπατε θέλουμε να πάμε στο 3% αλλά ότι καν στο 2% δεν είμαστε ακόμα για, την, για τις επενδύσεις στην έρευνα. Αν πετυχαίναμε το στόχο 3% θα αρκούσε σε σχέση με τις άλλες χώρες Ινδία, Κίνα και Αμερική. Οι ανεπαρκείς λοιπόν πόροι και κονδύλια για να φέρουμε στην έρευνα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθούν συντονισμένα εφόσον έχουν τον ίδιο στόχο. Η ευχή μου είναι, σε σχέση με αυτή την ευκίνητη δομή που αναφέρατε, το κόστος ποιο θα είναι το λειτουργικό κόστος και ποιο θα είναι το κόστος των προγραμμάτων για να έχουμε μια καλή ισορροπία για να δούμε αν είναι χρήσιμη μια τέτοια δομή ή όχι. Πρόεδρος, τελευταία ομιλητρία, συνάδελφος Τικάου. Παρακαλώ. Ε, μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Αν ο κύριος ε, Σούρμαν θέλει να τα απαντήσει όλα. Κυρία Τικάου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο ερωτήματα. Μία παρατήρηση μάλλον και μία ερώτηση. Πολύ σύντομα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει πάρα πολλά κονδύλια στην έρευνα. Τα οποία ήταν όλα επιτυχή. Έχουμε λοιπόν τώρα διαθέσει πολλά, πολλές πιστώσεις για την έρευνα, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε επενδύσει αρκετά σε έναν άλλο τομέα. Στον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας. Ε, το οποίο θα μας επέτρεπε να μετατρέψουμε τα ερευνητικά αποτελέσματα σε χειροπιαστά προϊόντα στην αγορά τα οποία συνεχεία θα μπορούν να αποδώσουν ένα οικονομικό όφελος. Εδώ δεν τα έχουμε καταφέρει καλά. Ρωτώ λοιπόν εάν μία από τις στρατηγικές από τους στρατηγικούς στόχους του Ινστιτούτου είναι να προωθήσει ε, πρωτοβουλίες ε, και ενοτομίες στον τομέα της ε, ενέργειας. Και είμαι πρόθυμη και θέλω επίσης να σας ρωτήσω στον τομέα της καινοτομίας τι, θα, τι στόχους έχετε για την αηφόρο ανάπτυξη και τις αηφόρους ενεργειακές πηγές. Είπατε ότι θα διαλέξετε μέχρι το Δεκέμβριο θα επιλέξετε τρεις καινοτομικές κοινότητες και θα θέλαμε να ξέρετε ποια θα είναι τα θέματα αυτών των κοινοτήτων και πώς θα διαθέσετε τις επενδύσεις για τις κοινότητες αυτές, ειδικά στην έρευνα για την, ενέργεια και την ενεργειακή απόδοση. Θα πρέπει να απαντήσετε τηλεγραφικά, λέει ο Πρόεδρος. Ε, τι να κάνετε. Μου φτάνει, μου φτάνει, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, πάρα πολλές ερωτήσεις και σας ευχαριστώ θερμά, επειδή ήταν πολύ επίκαιρες και πολύ ενδιαφέρουσες. Θα σας ε, παρουσιάσω δύο οριακές προδιαγραφές, ένα πλαίσιο δηλαδή που, θα, που εξηγεί ε, την ε, προσέγγιση μου. Καταρχάς η επιτυχία βασίζεται στην επιτυχία. Πρώτα λοιπόν πρέπει να σημειώσεις μία επιτυχία για να προχωρήσεις στις επόμενες. Εφόσον λοιπόν ζητάτε μεγαλύτερη ορατότητα, μεγαλύτερη διάβια όσον αφορά τις καινοτομίες, θα πρέπει πρώτα να φτάσουμε στο επίπεδο επιλογής των ΚΙΚΣ και εν συνεχεία να, δείξε, να δείξουμε σε όλους ε, τι επιτυχίες έχω στο νου μου να ε, προβάλλω και πώς μπορούμε να δικαιολογήσουμε τα χρήματα και τις πιστώσεις. Ε, ένας άλλος, μία άλλη προσέγγιση δική μου είναι ότι δεν θέλουμε να κάνουμε τα πάντα για τους πάντες. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, διότι υπάρχει τέση να πούμε ότι τώρα που έχουμε αυτό το Ινστιτούτο ας καλύψουν θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, θέματα εκπαίδευσης, θέματα ε, κοινωνικών ε, επιπτώσεων, ε, πώς ας πούμε θα προωθήσουμε την έρευνα στην κοινωνία. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία και σημαντικά θέματα, αλλά εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη δουλειά να κάνουμε, η οποία ε, δεν καλύπτει όλα αυτά τα επιμέρους θέματα. Θα είμαι λοιπόν πολύ ε, ειλικρινής. Βεβαίως ε, θα δώσουμε σημασία σε αυτές τις πτυχές, αλλά δεν είναι ο βασικός μας στόχος. Τώρα, επιστήμη στην κοινωνία, οπωσδήποτε πρέπει να την προωθήσουμε. Επιστημονικές έρευνες, παρουσία της επιστήμης στην κοινωνία. Όταν τώρα, όπως ρώτησε η κυρία Καλβάλιο, ε, ασχολούμεσα με τις νέες μορφές της τεχνολογίας βεβαίως με ενδιαφέρει και παρακολουθώ τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα και πολλές φορές όταν πηγαίνω στις ΗΠΑ απελπίζουμε όταν βλέπω τι γίνεται στην Αφρική, στην Νότια Αμερική για το κρασί και στο γεωργικό τομέα γενικά. Ε, λέω γιατί η Ευρώπη δεν, δεν ηγείται αυτών των ερευνών, αυτών των καινοτομιών όταν τόσα πράγματα σημειώνονται σε άλλες υπήρους. Αλλά σας είπα, δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα. Είπαμε ότι στον επόμενο γύρο θα καλύψουμε υγεία και διατροφή, υγεία και τρόφιμα. Τρόφιμα, διατροφή και υγεία που πιστεύω έχει θεμελιώδη σημασία τον πληθυσμό μας. Και θέλω να πω ε, λίγα λόγια για, τα, για τους οργανισμούς και τα Ινστιτούτα Κλειδί και τους άλλους ε, συναφείς οργανισμούς. Οι λεγόμενοι key showstoppers, δηλαδή τα Ινστιτούτα Κλειδιά, τα Ινστιτούτα Πρωτοπορίας, οδηγούν το δρόμο. Εμείς ε, προήλθαμε από μια κατάσταση όπου θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι σκορ θα επιτύχουμε. Περισσότερα χρήματα, ναι. Αυτό είναι μια σωστή και δικαιολογημένη ερώτηση. Πιστεύω ότι τα αποτελέσματά μας θα δικαιολογήσουν την χρηματοδότησή μας. Τα, IPR, τα πνευματικά δικαιώματα, δεν είναι ένα θέμα κλειδί για μας Όταν δείτε ε, τι σημασία έχει το πρόβλημα των ε, πνευματικών δικαιωμάτων στην ατζέντα όταν συζητάει κανείς ε, στην Ινδία ή στην Κίνα διάφορα θέματα θα δείτε είναι τελευταίο στην ατζέντα. είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα και όταν προκύψει ένα θέμα IPR τότε θα πρέπει να πας στον συνομιλητή και να του πεις κοίταξε αυτό και αυτό συνέβη θα το λύσουμε επιτόπου, ad hoc, επιτόπου εδώ και τώρα δεν μπορούμε να το προκαταλάβουμε Τώρα, η, επαναλαμβάνω ότι η διεθνή η παγκόσμια διάσταση είναι βεβαίως πάντοτε παρούσα, αλλά εγώ προτιμώ να προβάλλω την ευρωπαϊκή θέση. Το σφαιρικό, το παγκόσμιο, πάντα μας απασχολεί. Αλλά ε, να προβάλλουμε την Ευρώπη, να προχωρήσουμε εμεί η Ευρώπη. Γι' αυτό θέλουμε να αναλάβουμε και ε, ηγετικό ρόλο στην κοινοτομία και στην τεχνολογία. Και καταλήγοντας πρόεδρε, θέλω να πω ότι Θέλουμε να συγκεράσουμε τα κέντρα αριστείας τα οποία και γεωγραφικά και ε, επί του περιεχομένου είναι πάρα πολύ κοντά το ένα στο άλλο και όλοι οι άλλοι φορείς μέσα στο δίκτυο αυτό θα υποφεληθούν. Διότι από τη στιγμή που θα συγκεράσουμε και θα δημιουργήσουμε ένα ε, ε, πολύ δραστήριο δίκτυο ε, συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων φορέων της καινοτομίας και της τεχνολογίας ε, θα ξεπεράσουμε τα εθνικά σύνορα. Εάν δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τα εθνικά σύνορα θα συμβεί ακριβώς το ίδιο ε, με αυτό το οποίο έγινε στη δική μου χώρα, το Βέλγιο, όπως και στη Γερμανία, στεγανά. Στεγανά και απομονωμένες κοινότητες έρευνας και τεχνολογίας ε, και καινοτομίας. Γι' αυτό λοιπόν, ε, συνεργασία, συγκερασμός. Ελπίζω να, να απάντησα γενικά βεβαίως. Ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που διαθέσατε, για τον ενθουσιασμό με τον οποίο μας μιλήσατε. Είμαι βέβαιος ότι κερδίσατε την υποστήριξη των ακροατών σας και θα σας ε, θα έχουμε την ευκαιρία σίγουρα τα επόμενα χρόνια να σας βλέπουμε τακτικά. Εύχομαι ε, καλή επιτυχία στα, ε, στο έργο σας και λέω όπως είπε και ο Ομπάμα just do it, κάντο, κάντο, φτιάξτε το, κάντο. We'll do it. And we're on time,